το βάθος, αλλά ελπίζω να τους εντυπωσιάσουμε αργότερα. Λοιπόν, θα έχουμε κάποιον εκπρόσωπο από την Υπηρεσία Προσφύγων των Ηνωμένων Εθνών και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εμείς ζητήσαμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή επί τη βάση της πρωτοβουλίας της Αυστριακής να δημιουργήσουμε ένα αντίστοιχο σύστημα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ε, πρόκειται για το πρόγραμμα Safe Lives στο Αυστριακό. Τα είχαμε συζητήσει σε ένα πρώτο επίπεδο. Μια τελευταία συνάντηση ε, που θα οδηγούσε σε ένα δεύτερο φόρουμ ακυρώθηκε. Και τώρα το θέμα παραμένει να προσπαθήσουμε να πάρουμε μια καλύτερη ιδέα η κυρία Φιλίπα Κάντλερ θα μας μιλήσει για τις ε, επαφές σε υπουργικό επίπεδο σε σχέση με την επανεγκατάσταση και άλλες ε, μορφές ε, υποδοχής που συζητήθηκαν στη Γενέβη, στη το Δεκέμβριο του 2014. Θα δώσω πρώτα λοιπόν τον λόγο στην κυρία Κάντλερ από το Ευρωπαϊκό Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες. Ακόμα και χωρίς PowerPoint, αν αρχίσει να δουλεύει τόσο το καλύτερο. Έχετε το λόγο λοιπόν. Και μετά θα δώσω το λόγο στον κύριο Λογάν Μισελ που είναι εκπρόσωπος της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων. Σας ευχαριστώ πολύ. Λέγομαι Φιλίπα Κάντλερ, Εργάζομαι για την υπηρεσία του Ηνωμένων Εθνών για τους πρόσφυγες εδώ στις Βρυξέλλες. Σας ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας. Δύο είναι τα θέματα στα οποία μου ζητήσατε να κάνω τα σχόλιά μου. Καταρχάς για την συνάντηση τον Δεκέμβριο του 2014 για την προστασία στη θάλασσα των προσφύγων και δεύτερον η διάσκεψη που έγινε επίσης το Δεκέμβριο στη Γενέβη για τις ε, αναλήψεις υποχρεώσεων από πλευράς των κρατών μελών σε σχέση με τις επανεγκαταστάσεις προσφύγων. Μια καταγραφή των αναγκών δηλαδή, των προσώπων με τα οποία ασχολούμεθα εμείς σαν υπηρεσία προσφύγων. Οι περισσότεροι γνωρίζετε τα βασικά στοιχεία, αλλά στο τέλος του 2014 είχαμε 15 εκατομμύρια εκτοπισμένους βίαια και πρόσφυγες και ανθρώπους οι οποίοι είχαν εκτοπιστεί σε εσωτερικό επίπεδο, στο εσωτερικό των χωρών τους. Και αυτό περιλαμβάνει ε, κρίσεις όπως η Συρία με 3,8 εκατομμύρια πρόσφυγες, ιδιαίτερα στις γειτονικές χώρες της Συρίας, αλλά και στην Αίγυπτο και στη Βόρεια Αφρική. 7,6 επίσης εκτοπισμένους Σύρους, οι οποίοι παραμένουν εκτοπισμένοι σε εσωτερικό επίπεδο όμως. Um, perhaps also to note that um, at, by the end of 2014, non-industrialized countries οι μη βιομηχανοποιημένες χώρες ε, υποδέχθηκαν περίπου το 90% των προσφύγων στον κόσμο. Αλλά βέβαια ε, και στην Ευρώπη είδαμε έναν αριθμό αυξανόμενο των ανθρώπων που φτάνουν στην Ευρώπη. Για το 2014 έχουμε 600 κάτι χιλιάδες ε, που ζήτησαν άσυλο στις 28 χώρες ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, πάνω από 400.000 αφορούν αποκλειστικά χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ οι υπόλοιποι 200 κάτι αφορούν και τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης. Οι βασικές εθνικότητες αυτών οι οποίοι αιτούνται ασύλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση περιλαμβάνουν φυσικά πολίτες της Συρίας που είναι οι περισσότεροι αλλά και Ιρακινούς, Αφγανούς κτλ. Αυτές είναι οι τάσεις και έχουμε επίσης διαβάσει στον τύπο πολλά και για κατοίκους της Ερυθρέας οι οποίοι προσπαθούν να περάσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να υπογραμμίσουμε επίσης ότι η Σουηδία και η Γερμανία έχουν δεχθεί το 46% των αιτήσεων αυτών έχουν υπάρξει επίσης και πάρα πολλές συζητήσεις και για τις αφήξεις μεσοθαλασσίων μέσων. Υπήρξε μια τεράστια αύξηση το 2014 στις θαλάσσιες αφήξεις, πάνω από 218.000 που διέσχισαν ε, την ε, ε, Μεσόγειο και το μεγαλύτερο ποσοστό πήγε στην Ιταλία. Αυτό που σημειώνουμε με ανησυχία είναι ότι οι μισοί από αυτούς προέρχονται από χώρες οι οποίες παράγουν ε, πρόσφυγες συστηματικά όπως και η Ερυθρέα. Αυτή η αυξανόμενη τάση ε, άφηξης από, θαλάσσας, ε, επιβεβαιώνεται μέχρι τώρα και για το 2015 3.500 έφτασαν στην Ιταλία ενώ το αντίστοιχο χρονικό διάστημα ήταν 2.171. 62% αύξηση δηλαδή στις αφήξεις στην Ιταλία ε, μόνο και μόνο για τους δύο πρώτους μήνες. Το 2014 τώρα παρά τις προσπάθειες οι οποίες έγιναν από πλευράς της Ιταλίας, της επιχείρησης Mare Nostrum, ε, υπήρξαν δυστυχώς 3.500 νεκροί ή αγνοούμενοι, 370 ε, αντίστοιχες περιπτώσεις δυστυχώς αναφέρθηκαν μέχρι τώρα και για το 2015. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με τους αριθμούς που είχαμε το 2014 όπου τους πρώτους μήνες είχαμε μόνο 12 που είχαν χάσει τη ζωή τους. Υπάρχει μια μεγάλη δηλαδή αλλαγή. Βέβαια αυτές είναι πρώτες εκτιμήσεις, είναι πάρα πολύ δύσκολο με βεβαιότητα να αναφερθούμε στους αριθμούς των ανθρώπων οι οποίοι εντάσσονται στις προαναφερθήσεις κατηγορίες. Τώρα ας περάσουμε λίγο στο πρώτο τμήμα της παρουσίασής μου, τον διάλογο δηλαδή ε, της ε, Υπηρεσίας των Ηνωμένων Εθνών για την Συνδρομή στην Θάλασσα. Ξεκίνησε ένας διάλογος για τα βασικά θέματα προστασίας. Το 12 τέθηκαν θέματα θρησκευτικά, το 13 εσωτερικοί εκτοπισμοί, αλλά βλέποντας ότι αυξάνεται ο αριθμός των ανθρώπων που κάνουν επικίνδυνες θαλάσσιες διαδρομές, το 2014 ασχοληθήκαμε με ε, τις θαλάσσιες μεταφορές των προσφύγων. Οι άνθρωποι που καταφεύγουν σε τέτοιες ε, διαδικασίες φυσικά εντάσσονται στην κατηγορία των ατόμων που ενδιαφέρουν την υπηρεσία μας. Δεν έχουμε φτάσει ακόμα σε ένα τελικό συμπέρασμα, έχουμε, είμαστε σε φάση μιας αρχικής συζήτησης. Υπήρξαν συζητήσεις ανάμεσα σε 88 χώρες, υπήρξαν εμπειρογνώμονες, πανεπιστημιακοί και φυσικά μη κυβερνητικέ οργανώσεις. 400 άτομα πήραν μέρος στον διάλογο που δείχνει τον τεράστιο ενδιαφέρον το οποίο υπάρχει για τη συνδρομή στην θάλασσα. Ε, ταυτόχρονα με την οργάνωση του διαλόγου αρκετές οργανώσεις μεταξύ των οποίων και η δική μας αλλά και η Διεθνής Οργάνωση Μετανάστευσης, η Διεθνής Ναυτιλιακή Οργάνωση, η ύπατη αρμοστία για τα ανθρώπινα δικαιώματα ε, έκαναν μια κοινή δήλωση ζητώντας από όλα τα κράτη να αντιμετωπίσουν τις ρίζες που είναι πίσω από τις θαλάσσιες αυτές μετακινήσεις. Και τέθηκαν αρκετά θέματα στα πλαίσια αυτής της συνάντησης μεταξύ των οποίων το θέμα της απόβασης ε, των παρανόμων μεταναστών, όπως επίσης και το θέμα της κατανομής των ευθυνών, το θέμα της κατανομής του βάρους μέσω της διεθνούς συνεργασίας κτλ. κτλ. Ε, τέλος καταλήξαμε στο ότι υπάρχει μια συνένεση σχετικά με τα θέματα πρόληψης. Συμφωνήσαμε επίσης στο ότι οι μονομερείς ενέργειες δεν πρόκειται να σταματήσουν τις διαδικασίες αυτές και υπήρξε και μια ισχυρή εδώ αναφορά στην ανάγκη για δημιουργία επαφών όχι μόνο για την μετανάστευση αλλά για την πλευρά την αναπτυξιακή. Υπήρξαν και άλλες ε, συζητήσεις για την κατανόηση και την εξήγηση ε, των χωρών προέλευσης και των χωρών υποδοχής. Ε, προσπαθήσαμε ε, να δούμε τον λόγο για τον οποίο φεύγει ο κόσμος, εγκαταλείπει τις χώρες του και φυσικά ε, οι περισσότερες από τις κρίσεις αυτές οφείλονται σε πολιτικούς βέβαια λόγους και αν επιληθούν οι πολιτικοί αυτοί λόγοι μπορεί να μειωθούν οι αριθμοί. Αλλά παρόλα αυτά απαιτούνται περισσότερες προσπάθειες για να αποτρέψουμε την εκμετάλλευση αυτών των ανθρώπων από το οργανωμένο έγκλημα. Τέθηκε επίσης και το θέμα για τα νομικά εναλλακτικά μέτρα. Ένας από τους καλύτερους τρόπους για να προλάβει κανείς τέτοιου είδους μεταφορές θαλάσσιες ε, είναι να αυξήσουμε την ε, δυνατότητα οι άνθρωποι αυτοί να πηγαίνουν σε ασφαλείς περιοχές και να μένουν εκεί και να μην εξαναγκάζονται να διακινδυνεύσουν το πέρασμα της ε, θαλάσσιας περιοχής. Τέθηκε επίσης και το θέμα της αναζήτησης και ε, συνδρομής ιδιαίτερα σε περιοχές της Μεσογείου και την ανάγκη που υπάρχει για την έρευνα και διάσωση στις περιοχές αυτές. Όπως επίσης και πρακτικά θέματα στην περίπτωση κατά την οποία τα πρόσωπα αυτά ε, διασωθούν. Ε, όλα αυτά λοιπόν εξηγούν εν πολλής το σημερινό αυτό κοινωνικό φαινόμενο και εμεί πρέπει να κάνουμε ένα βήμα προ τα μπρο. Γι' αυτό λοιπόν και χαιρόμαστε πάρα πολύ για τι πρωτοβουλίε που λαμβάνουν χώρα στην Ευρώπη, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για παράδειγμα. Η προσέγγιση για τη μετανάστευση είναι ένα θετικό βήμα προ τα μπρο, όπω επίση και η έκθεση πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που εξετάζει την κατάσταση στη Μεσόγειο και επιβεβαιώνει και την ανάγκη αυτή για μια πιο σφαιρική προσέγγιση και αντιμετώπιση. η παρουσίασή μου PowerPoint δεν λειτουργεί από ό,τι φαίνεται. Σας είπα ήδη πάντως ότι συζητάμε σε επίπεδο είπα της ε, αρμοστίας για την ε, επανεκατάσταση ότι δουλεύουμε πάνω στη δικιά μας προσέγγιση για την πρωτοβουλία κεντρικής Μεσογείου και νομίζω ότι έχετε και εσείς τεκμηρίωση. Σας δώσαμε δηλαδή εν ώψη αυτής της συνάντησης. Συνεχίζουμε πάντως τις συνομιλίες μας και με τους πλειοκτήτες που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία διάσωσης στη θάλασσα. Η υπηρεσία μας έχει αναλάβει επίσης να παρακολουθήσει και το πρόγραμμα δράσης που σκοπεύει να ξεκαθαρίσει κάπως το ρόλο που παίζουν οι διεθνείς οργανώσεις για την μετανάστευση και η υπηρεσία μας για τους πρόσφυγες. Ήδη στο Λονδίνο υπάρχει μια συνάντηση για τους μετανάστες και πρόσφυγες οι οποίοι ταξιδεύουν ε, με πρόχειρα σκάφη που δεν είναι ασφαλή στη Μεσόγειο. Θα είναι και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η δικιά μας υπηρεσία φυσικά. Και άλλες υπηρεσίες του ΟΙΕ επίσης. Η συνεργασία τώρα με την κοινωνία των πολιτών και τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις σε διάφορες περιοχές κλειδί. Και αυτό υπογραμμίζεται ότι είναι ένα σημαντικό τομέα που πρέπει να παρακολουθούμε. Κυρίως πρέπει να δούμε τι πληροφορίες μπορούμε να έχουμε από μη κυβερνητικέ οργανώσεις που δουλεύουν σε αυτές τις περιοχές για να μπορούμε να αναλύουμε τα δεδομένα και να μπορούμε να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα για τις διαδρομές που ακολουθούν οι άνθρωποι που μετακινούνται και από ποια περιοχή προς ποια περιοχή. Έχουμε μια γραμματεία στην Αϊρόμπη, για παράδειγμα, που εξετάζει ακριβώς τέτοιου είδους θέματα. Στήριξη των ε, μεταναστών τώρα σε χώρες που βρίσκονται σε κρίση. Είναι και αυτό κάτι που θα παρακολουθήσουμε μετά το διάλογο της υπατής αρμοστίας. Κάτι στο οποίο θα αναφερθώ αργότερα είναι ότι θέλουμε να βρούμε και άλλους δρόμους για να βοηθήσουμε ανθρωπιστικά τους ανθρώπους αυτούς. Υπάρχουν δράσεις που προτείνουμε βάσει του διαλόγου της ΥΠΑ Αρμοστίας για την προστασία στη θάλασσα. Κάποιοι από εσά στην αίθουσα εδώ σίγουρα συμμετείχατε στο διάλογο αυτό. Σίγουρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμμετείχε, το ξέρω. Τώρα επιτρέψτε μου να πάω λίγο στις περιφερειακές πρωτοβουλίες που δεν είναι άμεσα συνδεδεμένες με το διάλογο της ΥΠΑ της Αρμοστίας. Είναι η πρωτοβουλία για την Μεσόγειο. Α, βλέπω ότι έχουμε τώρα την παρουσίαση PowerPoint, αλλά πρέπει να προχωρήσουν οι διαφάνειες. Ναι, εδώ είμαστε. Μα όλοι έτσι κι αλλιώς έχουν την παρουσίαση. Η πρωτοβουλία λοιπόν για την Κεντρική Μεσόγειο είναι μια πρωτοβουλία της ΥΠΑ της Αρμοστίας με διάφορες υπηρεσίες προστασίας για να δούμε τι έχουμε να συστήσουμε για την περιοχή αυτή της Μεσογείου. Ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2013 μετά την τραγωδία στη Λαμπετούζα και προτείνουμε έτσι 12 δράσεις εξετάζοντας τις χώρες προέλευσης, εξετάζοντας τις χώρες transit και εξετάζοντας και την κατάληξη στις ευρωπαϊκές χώρες. Για δράσεις και συστάσεις τώρα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στα πλαίσια αυτής της πρωτοβουλίας εξετάσαμε και αυτό το θέμα και επικεντρωνόμαστε σε δράσεις διάσωσης στη θάλασσα. Και εμείς και άλλοι εταίροι δίνουν πολύ μεγάλη σημασία σε αυτό. Ξέρουμε τι έχει κάνει η Ιταλία και πώς αναγκάστηκε να μειώσει τέτοιες δράσεις πρόσφατα. Βέβαια όλα αυτά έχουν να κάνουν και με τα νούμερα. Πόσοι δηλαδή διασχίζουν τη Μεσόγειο για να φτάσουν στις χώρες μας και πόσους θανάτους έχουμε στη θάλασσα το 2015 περισσότερους από ό,τι είχαμε την αντίστοιχη περίοδο το 2014. Η έκκληση αυτή αναγνωρίζει ότι παρόλο που η Frontex έχει τη δράση τρίτων, δεν έχει την εντολή ούτε τους πόρους για να προβεί σε διάσωση στη θάλασσα. Ένα άλλο σημείο δράσης που προτείνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι να μπορούμε να προβλέψουμε πόσοι θα διασωθούν από εμπορικά σκάφη. Μπορεί στο παρελθόν να μην ήταν πρόβλημα αυτό καθ' αυτό, αλλά τουλάχιστον πρόσφατα, πιο παλιό όμως ήταν. Και έχουμε αναπτύξει και νέο υλικό. Το πακέτο απάντησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν φτάνουν κάποιοι δηλαδή σε μια χώρα μέλος, πώς αντιδρούμε. Εδώ επικεντρωνόμαστε πολύ στο θέμα της ταυτοποίησης των ατόμων, ότι μπορεί να χρειάζονται διεθνή προστασία ή όχι και προσπαθούμε να βρούμε τι άλλες λύσεις υπάρχουν αν δεν εμπίπτουν στην κατηγορία αυτή των ατόμων που χρειάζονται διεθνή προστασία. Μπορεί να υπάρχουν κάποιοι που έχουν ανάγκη από ιατρική περίθαλψη, για παράδειγμα θέλουμε όταν φτάνουν στις χώρες μας να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις ανάγκες τους αυτές κατάλληλα. Η ταυτοποίηση είναι στοιχείο κλειδί σε αυτό το στάδιο. Γίνονται διάφορες συζητήσεις για την ασφάλεια τελευταία και η άποψη της είπα της αρμοστής για τους πρόσφυγες είναι ότι ακριβώς η αναγνώριση αυτή πρέπει να γίνεται μόλις φτάνουν, να ξέρουμε ποιοι είναι, να έχουμε το προφίλ τους. Καταγραφή σε ένα μητρό, τι συμβουλές ε, ενδεχομένω <coughs> πρέπει να τους δώσουμε. Εμείς συνεργαζόμαστε για να εφαρμοστεί ε, ο κανονισμός του Δουβλίνου. Στην Ευρώπη, αλλά και όχι μόνο, έχουμε κανόνες που βοηθούν τους ανθρώπους που φτάνουν αυτοί, οι οποίοι για παράδειγμα μπορεί να έχουν συγγενείς σε άλλες χώρες μέλη από, από αυτήν στην οποία φτάνουν μπορούν να χρησιμοποιηθούν τέτοια επιχειρήματα για να διευκολυνθεί η μετακίνηση των ατόμων αυτών προς άλλες χώρες μέλη. Επίσης πρέπει να δούμε η ρήτρα διακριτικής μεταχείρισης πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Σύριοι ή από την Ερυθρέα, για παράδειγμα, που ΣΥΡΙ η πρόταση αυτή είναι οι λύσεις ένταξη στη χώρα στην οποία βρίσκονται, επανένωση με μέλη της οικογένειάς τους εφόσον αυτό προκύπτει σε άλλη χώρα μέλος, αλλά και πέρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αν έχουν συγγενείς σε άλλες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην Ευρώπη ή αλλού. Γιατί κάποιοι μπορεί να έχουν ένα σύζυγο στις ΗΠΑ ή στον Καναδά. Οπότε θα ήταν μια λύση η μετακίνησή τους προς τα και αλλιώς οι αριθμοί δεν είναι πολύ μεγάλοι, αλλά για όσους προκύπτει αυτό είναι καλό να μπορούμε να τους προσφέρουμε αυτή τη λύση. Τέλος, η επιστροφή για αυτούς οι οποίοι δεν χρήζουν διεθνούς προστασίας. Η ύπατη αρμοστία δεν έχει αντίρρηση. Εφόσον δεν υπάρχει άλλος νόμιμος τρόπος για να παραμείνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τότε πρέπει να προβούμε στην επιστροφή με αξιοπρέπεια, κατά ανθρώπινες συνθήκες, σε θελοντική βάση κατά προτίμηση, και γι' αυτό και στηρίζουμε τα προγράμματα για την ε, επιβοηθούμενη επιστροφή σε θελοντική βάση. Αυτά λοιπόν προτείνουμε λίγο πολύ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όσον αφορά την πρωτοβουλία για την Κεντρική Μεσόγειο. Συνεργαζόμαστε και με τις χώρες πρώτου ασύλου για να υπάρχουν βιώσιμα συστήματα ασύλου, κάτι το οποίο έχει κάνει η Πατιαρμοστία και σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και συνεχίζει να κάνει πρόσβαση σε βιώσιμες λύσεις, για ευκαιρίες, για αυτονομία, για κατάρτιση, για σε βάση επιστροφή στις χώρες τους όπου αυτό προκύπτει, επανεκατάσταση ή άλλες λύσεις αν έχουν συγγενείς αλλού. Και με τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχουμε αναπτύξει και μία εκστρατεία ενημέρωσης στη Σομαλία και την Ερυθρέα και το κέντρο της Αφρικής και το Σουδάν προκειμένου να επικεντρωθούμε στα μηνύματα που πρέπει να στείλουμε. Δηλαδή ότι το ταξίδι μπορεί να είναι επικίνδυνο, ότι υπάρχουν και άλλες νομικές λύσεις. Θέλουμε δηλαδή να παρουσιάσουμε στους ανθρώπους αυτούς τι εναλλακτικέ λύσεις έχουν αντί να έρθουν στην Ευρώπη. Επανεγκατάσταση και μετεγκατάσταση. Το τρίτο σκέλος έχει να κάνει με τις χώρες προέλευσης. Έχουμε και εκεί δραστηριότητες για την υπατερμοστία ε, βέβαια είναι περιορισμένες, αλλά συνεργαζόμαστε με οργανώσεις εταίρους που έχουμε εκεί, σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα, σχετικά με προγράμματα ανακούφισης σε συνεργασία με το αναπτυξιακό πρόγραμμα το ΟΗΕ και προγράμματα ένταξης για τα άτομα που επιστρέφουν στις χώρες τους. Αυτά όσον αφορά την πρωτοβουλία και την κεντρική Μεσόγειο. Έρχομαι τώρα στη δεύτερη πτυχή, το δεύτερο πράγμα για το οποίο μου ζητήσατε να σας μιλήσω σήμερα. Αυτό είναι η επανεκατάσταση. Resettlement. Νομίζω ότι συνδυάζεται πάρα πολύ καλά με τις πρωτοβουλίες που προτείνουμε στα πλαίσια της Κεντρικής Μεσογείου. Θέλουμε η επανεκατάσταση αυτή να ενισχυθεί. Αυτά είναι τα νούμερα, οι εκτιμήσεις δηλαδή της είπα της αρμοστίας 960.000 πρόσφυγες. Το 2014 είχαμε 94.000 εισδοχές σε διάφορες χώρες Η μεγαλύτερη χώρα βέβαια σε αυτή την περίπτωση που έχει πάρει τους περισσότερους δηλαδή είναι οι Ηνωμένε Πολιτείε, κάπου 60.000 κάθε χρόνο ως επανεκατάσταση. Είναι μεγάλη αναλογία αυτή. Δεν έχουμε στοιχεία για άλλες περιπτώσεις 71.000 έφυγαν πάντως το 2013 για επανεγκατάσταση, οι περισσότεροι προς την Ευρώπη. Ποιες είναι οι προτεραιότητές μας. Τα έχετε στο υλικό που σας έδωσα, δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες. Πάντως, η κύρια περίπτωση που αντιμετωπίζουμε σήμερα είναι η κατάσταση στη Συρία. Εδώ η επανεκατάσταση είναι η απάντηση που δίνουμε σε ένα μεγάλο βαθμό στην κατάσταση αυτή κρίσης που αντιμετωπίζουν οι Σύριοι πρόσφυγες. Από πλούρας επανεγκατάσταση, επίσης Έχουμε κάποια προφίλ προτεραιότητας που είναι πρώτα απ' όλα οι γυναίκες και τα κορίτσια που κινδυνεύουν όσοι έχουν βασανιστεί, άλλοι που χρειάζονται φυσική προστασία, αλλά και πρόσφυγε με άλλου είδους ανάγκες επειδή είναι ευάλωτοι. Τα προφίλ που επεξεργαζόμαστε τώρα για την επανεγκατάσταση πάντως κυρίως είναι όσοι έχουν επιβιώσει βασανιστήριων και όσοι χρήζουν φυσικής προστασίας. Υπήρξε και η υπουργική διάσκεψη στην Γενέβη. Συμμετείχαν 40 χώρες και η Διεθνής Οργάνωση για την Μετανάστευση και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήταν εκεί και άλλες οργανώσεις, 26 χώρες προσέφεραν 58.000 θέσεις περίπου και πάρα πολλές επίσης στις Ηνωμένε Πολιτείες. Πάνω από 80.000 συνολικά. Επιπλέον, έχουμε και άλλου είδους θεωρήσεις που έχουν δοθεί σε Σύριους, 12.000 συνολικά, με άλλου είδους εισδοχή. Και η Βραζιλία και η Γαλλία και η Γερμανία και η Ιρλανδία και η Ελβετία και το Ηνωμένο Βασίλειο με διαφορετικό τρόπο καθεμία υποδέχονται Σύριους πρόσφυγες. 19 ευρωπαϊκές χώρες επίσης έχουν προσφέρει βοήθεια, 15 από την Ευρωπαϊκή Ένωση, με 70.000 θέσεις απασχόλησης. Κάτι πολύ θετικό. Συγγνώμη, 37.000 θέσεις. 37.000 θέσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση, 30.000 ήταν από τη Γερμανία. Είναι ενδιαφέρον να συγκρίνει κανείς την περίπτωση της Γερμανίας με τις άλλες χώρες. Όπως σας είπα υπάρχουν και άλλου είδους προγράμματα από τη Γαλλία, την Ιρλανδία, έχουν ένα πρόγραμμα εισδοχών λόγω ανθρωπιστικών αναγκών και το Ηνωμένο Βασίλειο. Θα προχωρήσω γιατί μου είπαν ότι πρέπει να έχουμε χρόνο και για ερωτήσει. Να αναφερθώ επίση και στα συμπεράσματα του Συμβουλίου Δικαιοσύνη το Οκτωβρίου του 2014 που ζητάει από τα κράτη-μέλη να προσφέρουν θέσει επανεκατάσταση σε εθελοντική βάση όσο γίνεται πιο γρήγορα. Και αυτό είναι κάτι το οποίο στηρίζει πάρα πολύ η υπατιαρμοστία για τους πρόσφυγες άλλοι τρόποι εισδοχής τώρα που θα ήθελα να σας εξηγήσω. Μιλάμε εδώ πέρα για ανθρωπιστικές θεωρήσεις, για συστήματα χορηγίας. Η Γερμανία έχει ήδη προχωρήσει προς αυτή την κατεύθυνση και θα θέλαμε και άλλες χώρες να το κάνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να αποτελέσει μοντέλο και για άλλους. Υπάρχει επίσης η υποδοχή συγγενών πέρα από την οδηγία για την επανένωση οικογενειών. Πάλι και αυτό έχει να κάνει με ιδιωτικές χορηγίες. Υποτροφίες επίσης για φοιτητές, μαθητές, αλλά και βοήθεια για εργασία σε πρόσφυγες. Με κάποιες προϋποθέσεις βέβαια. Και το τελευταίο που θέλω να πω είναι η ένταξη. Χαιρόμαστε που συμμετέχουν περισσότερες χώρες στην επανεκατάσταση, αλλά οι χώρες πρέπει να είναι έτοιμες με βιώσιμα συστήματα για να μην μετακινούνται οι πρόσφυγες αυτές και μετά την επανεκατάσταση βρεθούν αλλού. Αυτά. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Όλοι έχετε λάβει την παρουσίαση αυτή, γι' αυτό θα σας ε, ζητούσα να είστε σύντομοι, έτσι ώστε να μπορέσουν να απαντηθούν όσο δυνατόν περισσότερες ερωτήσεις. Το δεύτερο μέρος της ενημέρωσης της υπατεσσαρκοστής προέρχεται από τον ε, Λοράν Μισελ, αλλά νομίζω πως αναφέρατε και εσείς στην έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας και είχαμε και έναν από τους ε, εισηγητές εδώ. Ο λόγος για τον οποίο ζητήσαμε αυτή την ενημέρωση είναι για να αποκτήσουμε μια πιο ε, σφαιρική και επικαιροποιημένη εικόνα για την κατάσταση. Τώρα, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κύριε Μισελ, θα μπορούσατε κι εσείς να μας κάνετε την δική σας παρουσίαση και να σας κάνουμε μετά ερωτήσεις. Ίσως λίγο σύντομα, έτσι να μας σκιαγραφίσετε την κατάσταση. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καταρχά πρωτού σας ενημερώσω για τα αποτελέσματα της ε, συνάντησή μα θα ήθελα να αντιδράσω σε κάποια πράγματα που είπε η κυρία Κάντλη για το τι πρέπει να γίνει και τι χρειάζεται. Θα ήθελα να αναφέρω κάτι για τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης. Χάρη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καταφέραμε ε, να έχουμε 20 εκατομμύρια επιπλέον ευρώ σε κονδύλια για έρευνα και διάσωση. Αλλά ας μην ξεχνάμε τι σημαίνει μια τέτοια επιχείρηση. Πριν από δύο εβδομάδες έχασαν τη ζωή τους περίπου 300 άτομα και πώς έγινε αυτό. Τους έβαλαν σε φουσκωτές βάρκες, τους έβαλαν το πιστόλι στον κρόταφο και τους έριξαν στη θάλασσα σε κύματα ύψους 5 μέτρων χωρίς σωσίβια. Μιλάμε για ανθρώπους από την υποσαχάρη Αφρική, οι οποίοι δεν έχουν δει θάλασσα ποτέ στη ζωή τους και φυσικά δεν ξέρουν κολύμπη. Γι' αυτό λοιπόν μην περιμένετε η Frontex να μπορέσει να διασώσει όλους αυτούς τους ανθρώπους. Χρειάζεται να αμυνθούμε γιατί πραγματικά τα μέσα ενημέρωσης μας άσκησαν τη κριτική. Δεν είμαστε μάγοι, δεν μπορούμε να βγάλουμε ένα ραβδί και να λύσουμε τα πάντα. Όταν φεύγει κόσμος από τη Λιβύη πάνω σε τέτοιες βάρκες, υπό τέτοιες συνθήκες, δεν μπορούμε να κάνουμε θαύματα. Τώρα, θα είμαι και σύντομος. Να σας ενημερώσω για τη συνάντηση της 25ης Νοεμβρίου. Ναι, είμαι σίγουρος πως θα είστε σύντομος και περιεκτικός, όπως ακριβώς ήσασταν μέχρι τώρα. Διότι τώρα μιλάμε για την κατάσταση στα κράτη-μέλη. Πιστεύω πως ε, εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατανοούμε απόλυτα τι κάνει η Frontex. Δεν είμαστε εδώ για να σας επιβλέψουμε. Αλλά αυτό που ζητάμε από εσάς είναι μία ενημέρωση για το τι νομίζετε πως ε, έγινε σε αυτές τις ε, συναντήσεις. Ναι, σίγουρα. Αλλά γεγονό είναι ότι τα μέσα ενημέρωση ε, μα ασκούν εντονότατη κριτική και σε εμά και στη Frontex και ε, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην Ευρωπαϊκή Ένωση εν γέννη. Λοιπόν, στη συνεδρίαση αυτή συζητήθηκαν τρία βασικά θέματα. Καταρχά, η κατάσταση με του πρόσφυγε, πώ μπορούμε να εφαρμόσουμε ε, μια καλύτερη ισορροπία ανάμεσα στα κράτη-μέλη όσον αφορά την απορρόφησή του. Έπειτα, κατάσταση και πώς ε, μπορούμε να ενεργοποιήσουμε έναν ενδοκινοτικό μηχανισμό μεταγκατάστασης σε περίοδους κρίσης και τρίτον ε, νομική αρρωγή για όσους αναζητούν ε, διεθνή προστασία. Συμπεράσματα τώρα. Καταρχάς, όλα τα κράτη-μέλη επέμειναν για τις δραστηριότητες μεταγκατάστασης και για μια καλύτερη ισορροπία και για τον εθελοντικό χαρακτήρα της μεταγκατάστασης. Έπειτα, νομικές οδοί. Τα περισσότερα κράτη-μέλη είναι της άποψης ότι το κυριότερο όπλο είναι η μεταγκατάσταση και δεν επιθυμούν η Ευρωπαϊκή Ένωση να επενδύσει σε άλλες νόμιμες μεθόδους εισόδου. Έγιναν οι συζητήσει για αυτήν την ε, θεώρηση, όμως δεν επιθυμούν η Ευρωπαϊκή Ένωση να νομοθετήσει για το θέμα αυτό. Η μεταγκατάσταση λοιπόν είναι η κύρια νομική οδός. Όσον αφορά τώρα την κατάσταση σχετικά με τη μεταγκατάσταση και την ε, ίση κατανομή της, υπήρξε μια συμφωνία να αρχίσει ένα πιλωτικό πρόγραμμα. Πρέπει καταρχάς να καθοριστεί ο αριθμός των ανθρώπων που μπορεί να δεχτεί η Ευρώπη και μετά να ε, ισχύσουν ορισμένα κριτήρια για την ε, διανομή αυτών των ανθρώπων. Τα κριτήρια θα μπορούσε να είναι ο ε, πληθυσμός της κάθε χώρας, το ΑΕΠ, ο αριθμός των ετούντων άσυλο στο παρελθόν και κάποια κράτη-μέλη ανέφεραν τα ποσοστά ανεργία. Διότι όταν ένα κράτο έχει υψηλό ποσοστό ανεργία, έχει πολύ μικρότερε πιθανότητε να εντάξει αυτόν τον πληθυσμό. Αυτά λοιπόν ήταν τα κριτήρια τα οποία συζητήθηκαν. Και βασισμένοι σε αυτά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υποβάλει μια πρόταση για ένα πιλωτικό πρόγραμμα και ελπίζουμε να συμμετέχουν όσο το δυνατόν περισσότερα κράτη-μέλη σε αυτό. Και να είμαι ειλικρινής μαζί σας δεν έχει νόημα να συμμετέχει η Γερμανία και η Σουηδία σε αυτό το πρόγραμμα, διότι ανέκαθεν είχαν τέτοιες, ε, τέτοια προγράμματα μεταγκατάσταση. Στόχο μα είναι τα κράτη-μέλη τα οποία μέχρι τώρα δεν είχαν ποτέ τέτοιο πρόγραμμα και θέλουμε να ε, συμμετέχουν λοιπόν αυτά. Επίση, ανέφερα τον εθελοντικό χαρακτήρα συμμετοχή. Αυτό που θέλουμε είναι να συμμετέχουν όσο το δυνατόν περισσότερα κράτη-μέλη σε αυτά τα προγράμματα και εκείνα που δεν συμμετέχουν τουλάχιστον να στηρίξουν τις επιχειρήσεις μετακατάστασης ε, και με αυτό εννοώ μέσω χρηματοδότησης, ε, μέσω διοικητικής υποστήριξης, μέσω βοήθεια στα κράτη τα οποία θα συμμετέχουν τη διαδικασία αυτή. Τέλος, όπως γνωρίζετε, τα κράτη-μέλη είναι αρκετά διστακτικά για την ε, μετεγκατάσταση. Φοβούνται ότι σε μεγάλες συγκεντρώσεις αριθμών και αυτό που γίνεται είναι να ε, δημιουργηθούν διάφορες εξαιρετικές ε, συνθήκες, ειδικέ περιπτώσεις όπου θα, μπορούν, θα μπορεί να πυροδοτείται μια τέτοια διαδικασία μετεγκατάστασης. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Προσπαθώ να αποκρισταλώσω τις απόψεις των κρατών μελών και φυσικά, ναι, όπως είπατε, υπάρχει μια μεγάλη ανισορροπία ανάμεσα στα κράτη-μέλη σχετικά με τη μετεγκατάσταση. Γι' αυτό λοιπόν ε, με ενδιαφέρε πάρα πολύ να μάθω την άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις προτάσεις αυτές. Φυσικά και έχουμε επίγνωση του τι συμβαίνει στη Frontex και το αναγνωρίζω αυτό. Τώρα, θα ήθελα να δώσω το λόγο στους, ε, στα μέλη μας για τις ερωτήσεις τους. Αρχίζουμε με τον κύριο Χαλέρ. Ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. Όπως ακούσαμε, η Σουηδία και η Γερμανία δέχονται σχεδόν το 50% των αιτήσεων για άσυλο. Και είναι αρκετά ενδιαφέρον αυτό, δεδομένου ότι αυτές οι χώρες απέχουν πάρα πολύ από τα σημεία εισόδου. Και είναι αδύνατο να φτάσει κάποιος σε αυτές τις χώρες χωρίς να περάσει από διάφορα άλλα κρατημέλη όπου θα έπρεπε κιόλα να γίνονται αυτές οι αιτήσει. Και αυτή η ανισορροπία νομίζω πως ε, μακροπρόθεσμα δεν θα μπορεί να είναι βιώσιμη. Ιδιαίτερα για ορισμένες σχετικά μικρές χώρες όπως η Σουηδία. Θα ήθελα λοιπόν να μάθω τις απόψεις σας σχετικά με το τι μπορούμε να κάνουμε. Ακόμα και αν είχαμε αυτό αυτό το ποσοστό διανομής ή αυτό τον μηχανισμό εξισορρόπησης, ε, μια που υπάρχει ελεύθερη μετακίνηση εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα μπορούσε κανείς να υποθέσει ότι οι άνθρωποι αυτοί θα προσπαθήσουν να μεταβούν σε αυτές τις χώρες, οι οποίες για τον ένα ή άλλο λόγο είναι πιο ελκυστικές για εκείνους, από ότι οι χώρες ε, στις οποίες ε, στάλησαν αρχικά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. έχουν ζητήσει πάρα πολύ το λόγο. Η Αναγκόμερ. Έχοντας επισκεφθεί την προηγούμενη εβδομάδα το κέντρο υποδοχής στην Βηρητό που εγγράφει 11.000 ε, πρόσφυγες τον μήνα. Πριν ένα εξάμεινο ήταν 50.000 το μήνα. Στο Λίβανο ε, μιλάμε για μια μικρή χώρα, το 1 τέταρτο της Ελβετίας και το 25% του πληθυσμού είναι πρόσφυγες από τον πόλεμο στη Συρία. Πάνω από ένα εκατομμύριο, ένα εκατομμύριο 200 χιλιάδες. Έχουν γίνει τεράστιες προσπάθειες για την υποδοχή τους και στην Ιορδανία ε, τον προηγούμενο μήνα επισκέφθηκα κέντρα υποδοχής στο Ιράκ ε, με Γεζιντή, Σαμπάκ και άλλες κοινότητες και είδα αυτά τα οποία κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα οποία δεν αρκούν. Δεν αρκούν φυσικά για να σταματήσει η σύγκρουση, δεν αρκούν ε, για να ε, σταματήσει η πίεση στους ίδιους τους πρόσφυγες. Υπάρχουν χώρες οι οποίες αναζητούν άλοθη για να μην μοιραστούν το δάρος, για να μην βοηθήσουν στην διάσωση στη θάλασσα, για να μην φανούν γενναιόδοροι και για να μην επενδύσουν σε ε, σωστούς δρόμους αντιμετώπισης του φαινομένου της μετανάστευσης. Δυστυχώς η κατάσταση με κάνει να ντρέπομαι. Η ερώτησή μου λοιπόν προς την εκπρόσωπο της ΥΠΑ της Αυμοστίας είναι η εξής. Αυτό το οποίο βρίσκω ιδιαίτερα ανησυχητικό και δεν μπορούμε να αντιμετωπίζουμε το παρόν πρόβλημα σε ανθρωπιστικό αποκλειστικά επίπεδο βέβαια γιατί υπάρχουν οι οποίοι δεν έχουν τη δυνατότητα να βοηθήσουν και χώρες που δεν έχουν τη δυνατότητα να βοηθήσουν αλλά βλέποντας τα δικά μας θέματα, τη δική μας ασφάλεια, τα δικά μας συμφέροντα. Γιατί να μην βοηθήσουμε σαν παράδειγμα σε σχέση με ε, την δημιουργία σχολικών δομών. Ε, στον Λίβανο ε, από τις 400.000 παιδιά που θα έπρεπε να πηγαίνουν σχολείο οι 320-330.000 δεν το κάνουν αυτό. Το θέμα δεν είναι λοιπόν να βοηθήσουμε τα παιδιά αυτά αργότερα να ανοικοδομήσουν την χώρα τους, αλλά να τα βοηθήσουμε τα παιδιά αυτά να μην γίνουν τρομοκράτες μεγαλώνοντας. Το ίδιο και στην Ιορδανία. Υπάρχουν άνθρωποι πρόσφυγες που θα μπορούσαν να διδάσκουν. Υπάρχουν κέντρα υποδοχής βέβαια στην Ιορδανία, τα οποία ελέγχονται καλύτερα. Στο Λίβανο δεν ελέγχονται οι άνθρωποι αυτοί αν κάναμε μία μικρή ε, έτσι και αλλιώς επένδυση επιπλέον θα βοηθούσαμε να δημιουργηθούν ε, σχολεία. Γιατί να μην το κάνουμε αυτό. Το ίδιο ισχύει και για το Βόρειο Ιράκ, για τη χριστιανική κοινότητα και την κοινότητα των Γεζιντή. Μία επιπλέον ερώτηση αφορά την Λιβύη. Εμείς όλα αυτά τα χρόνια είδαμε ότι αυτοί που έρχονται από τη Λιβύη με βάρκες δεν είναι Λίβοι, είναι Νιγηριανοί, Ερυθρέοι κτλ. Η κατάσταση έτσι όπως ε, είναι τώρα θα βλέπουμε όλο και περισσότερους ε, Λίβιους να έρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό φυσικά θα το εκμεταλλευτούν οι ε, εγκληματικές οργανώσεις θα στέλνουν κόσμο στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι εγκληματικές αυτές οργανώσεις για να κερδίσουν χρήμα. Συνεπώς λοιπόν πώς βλέπετε να εξελίσσεται η κατάσταση στη Λιβύη. Δεν νομίζω ότι πιστεύει κανείς ότι η κατάσταση θα βελτιωθεί. Ευχαριστώ αν. Όλοι οι συνάδελφοι είμαι σίγουρος ότι θα θέσουν πολύ σημαντικές ερωτήσεις αλλά θα ήθελα να σας ζητήσω παρακαλώ να μην μακριόρουμε. Λοιπόν, παρακαλώ προσπαθήστε να είστε συγκεκριμένοι και να περιοριστείτε σε λίγα σημεία. Ε, είναι σημαντική η έκθεση την οποία ετοιμάζουμε και θα τα συζητήσουμε αναλυτικά τα θέματα. Αυτά θα μπορέσετε να εκφραστείτε. Ε, σίγουρα αυτά ήταν πολύ σημαντικά, αλλά παρόλα αυτά θέλει λίγο προσοχή. Κύριε Χολμάιρ, καταρχάς θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και τους δύο για τις πιαρουσιάσεις σας. Τόσο την είπα τη Ηνωμένων των Εθνών, τόσο και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πραγματικά με έπεισε η ειλικρίνεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, γιατί αυτό που άκουσα είναι η σκληρή πραγματικότητα, σκληρή, βίαιη και άσχημη. Έχω τις εξής ερωτήσεις. Καταρχάς όσον αφορά τα στρατόπεδα των προσφύγων της ΥΠΑ Αρμοστίας του ΟΗΕ. Συμφωνώ απόλυτα με την Αναγκόμες με το ότι δεν μπορούμε να λύσουμε το πρόβλημα εάν δεν μπορούμε να δώσουμε με τον οποιονδήποτε τρόπο έστω μία προοπτική, μία ελπίδα σε αυτούς τους πρόσφυγες. Χρειάζονται ε, ε, αξιοπρεπείς όταν έχουν το ελάχιστο σε εγκαταστάσεις υγιεινής, το ελάχιστο σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη πρέπει να καταβάλουμε ως Ευρωπαίοι πολύ μεγάλη προσπάθεια και ειδικότερα εμείς οι Ευρωπαίοι, το τονίζω αυτό, να προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε την κατάσταση των ανθρώπων αυτών. Τουλάχιστον θα μπορούσαμε να ιδρύσουμε κάποια σχολεία για τα παιδιά που βρίσκονται σε, αυτά, σε αυτές τις εγκαταστάσεις προσφύγων. Διότι όλο ένα και αυξάνονται οι πρόσφυγες και μάλιστα υπάρχουν κάποια οι χώροι όπου είναι 20 ετών και φιλοξενούν πάρα πολύ μεγάλο αριθμό προσφύγων. Μπορείτε λοιπόν να φανταστείτε τι συμβαίνει εκεί, σε τι συνθήκες ε, ζουν οι πρόσφυγες αυτοί, πόσο άσχημες είναι αυτές οι συνθήκες. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν πάει ποτέ στο σχολείο γιατί μεγάλωσαν σε αυτά τα στρατόπεδα. Είναι πραγματικά χώροι με πάρα πολύ μεγάλα προβλήματα. Γι' αυτό λοιπόν θέλω να σας κάνω μία πάρα πολύ συγκεκριμένη ερώτηση για το τι γίνεται με τη χρηματοδότηση για δημιουργία σχολείων, για δημιουργία καλύτερων συνθήκων διαβίωσης, συνθήκων υγιεινής, πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα και ποια είναι τα συγκεκριμένα μέτρα τα οποία προτίθεται να λάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη. Επίση, η Frontex. Η Frontex δεν μπορεί να, να λύσει το πρόβλημα στη Λιβύη. Πώ θα αντιμετωπίσει το πρόβλημα στα σύνορα. Εδώ δεν φτάνετε μέχρι την ακτή της Λιβύης. Και η κυρία Μογκερίνη και τα κράτη-μέλη ανέφεραν το πρόβλημα και τη, την, τις ανθρώπινες ζωές που χάνονται, που τους πετάνε στη θάλασσα. Και πολλούς από αυτούς τους σκοτώνουν προτού καν φτάσουν στη θάλασσα, μέσα στη Σαχάρα. Αυτά τα πράγματα δεν συζητούνται τόσο πολύ, αλλά εκεί χάνουν τη ζωή τους τουλάχιστον όσοι χάνουν τη ζωή τους και στη θάλασσα. Γι' αυτό λοιπόν αυτές τις ερωτήσεις ήθελα να κάνω. Πρώτον, Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Frontex, ποια μέσα χρηματοδότησης υπάρχουν, τι προτίθεστε να κάνετε. Δεύτερον, υπάρχουν περαιτέρω σκέψεις για να ληφθεί κάποια στρατιωτική δράση όπως στην Σομαλία και τι διδάγματα έχουμε αντλήσει από αυτά που έχουν συμβεί στις ακτές της Λιβύης και στις, ε, βόρεια, της Βόρειας Αφρικής. Έπειτα, μηχανισμός ε, επανεγκατάστασης, ε, πώς συνεχίζει αυτό το πρόγραμμα. Πιστεύω πως εδώ χρειάζεται μεγαλύτερη συμμετοχή και ε, δικαίωμα επιλογής των κρατών μελών ε, των μηχανισμών που θα ακολουθήσει το καθένα και των μηχανισμών που μπορεί να ακολουθήσει το καθένα. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Ζήπελ έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Αυτό που θέλω να ρωτήσω εγώ την ύπατη αρμοστία αλλά και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όταν μιλάμε για τους καταβλισμούς ε, προσφύγων εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης Ποιος τους χρηματοδοτεί. Δεν είναι δυνατόν με τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι χώρες μέλη είναι διατεθειμένες να πληρώσουν. Δεν μπορούμε να καλύψουμε τους πρόσφυγες, να τους βοηθήσουμε, αλλά δεν μπορεί να μην κάνουμε και τίποτα μπορούμε να βοηθήσουμε, να δώσουμε μια προοπτική σε αυτούς οι οποίοι μπορεί να μην φεύγουν από πόλεμο, αλλά φεύγουν από δύσκολες καταστάσεις που τους καταδικάζουν στην ένδια. Αν μη τι άλλο, να δώσουμε μια προοπτική σε αυτούς τους ανθρώπους. Αλλιώς τα σημερινά προβλήματα θα συνεχιστούν. Δεν είναι δυνατόν να χτίζουμε τύχη για να μην βλέπουμε το τι συμβαίνει. Άρα το θέμα τίθεται περισσότερο στις χώρες μέλη για την επανεκατάσταση όμως, resettlement. Θέλω να ρωτήσω εκτός από την Επιτροπή, γιατί ξέρω και τα προβλήματα. Την είπατε αρμοστία για τους πρόσφυγες, θέλω να ρωτήσω. Βλέπετε δυνατότητα να δουλέψουμε πιο σκληρά στις χώρες μας, ώστε όλοι να συμμετάσχουμε στην επανεκατάσταση. Δεν συμβαίνει αυτό τώρα είναι μια θλιβερή κατάσταση. Μιλάμε για θεμελιώδη δικαιώματα, μιλάμε για το δικαίωμα στο άσυλο και μετά κάποιες χώρες λένε «Α, εμένα δεν με ενδιαφέρει, εγώ δεν θα συνεργαστώ». Υπάρχει περίπτωση να βελτιωθεί λοιπόν η κατάσταση και σταματάω εδώ γιατί ήδη έχουν τεθεί πολλά καλά ερωτήματα. Ευχαριστώ Μπριγκίτα, και ευχαριστώ που τήρησες τον χρόνο σου, λέει ο πρόεδρο. Προσπαθήστε να τηρείτε δύο λεπτά για να προλάβουμε να πάρουμε και απαντήσεις. Ο κύριος Κάρλος Κοέγιο τώρα έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ και για τις δύο παρουσιάσεις. Για την κυρία Κάντλερ, κάνατε κάποιες παρατηρήσεις για την αποστολή, την επιχείρηση τρίτων στην Μεσόγειο. Είπατε ότι δεν έχει τα απαιτούμενα μέσα και την εμβέλεια που απαιτείται. Θα συμφωνήσω μαζί σας, συμφωνώ την άποψη πολλών συναδέλφων, οι οποίοι πιστεύουν ότι είναι μια πάρα πολύ μικρή επιχείρηση σε σχέση με το μέγεθος της πρόκλησης. Θα ήθελα όμως τα σχόλιά σας σχετικά με την εντολή και την εμβέλεια. Είπατε ότι η επιχείρηση τρίτων δεν είναι υπεύθυνη για έρευνα και διάσωση. Κοιτάξτε, το Δεκέμβριο του 2013 εμείς εγκρίναμε έναν κανονισμό περιλαμβάνοντας και τις παρατηρήσεις της ΥΠΑ της Αρμοστίας και πολλών ΜΚΙΟ. Και καταφέραμε να πετύχουμε ένα συμβιβασμό ανάμεσα στο Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο εγκρίνοντας τον κανονισμό και δίδοντας συγκεκριμένες ε, ε, αποστολές στο Frontex. Αυτό δεν μπορούμε να το κάνουμε για τις εθνικές αποστολές. Όλες οι κυβερνήσεις πρέπει να έχουν τα δικά τους προγράμματα έρευνας και διάσωσης έτσι και αλλιώς. Όταν λέτε λοιπόν ότι δεν υπάρχει επαρκής εντολή και επαρκής εμβέλεια, είναι μεν σαφές, αλλά δημιουργούνται κάποιες περίεργες καταστάσεις. Ή δεν εφαρμόζεται ο κανονισμός, οπότε πρέπει να αναλάβουμε δράση, ή θα πρέπει να αλλάξουν τα πράγματα, να αλλάξει ο κανονισμός για να διορθωθεί η κατάσταση. Ευχαριστώ για τις ερωτήσεις σας. Κιέγγε. Ευχαριστώ. Οι ερωτήσεις που ήθελα να κάνω έχουν ήδη γίνει, αλλά ίσως να υπάρχουν κάποιες αμφιβολίες και απορίες που έχω σχετικά με τους χώρους υποδοχής εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ήθελα να μάθω για την ουσία του πράγματος μετά από τις εμπειρίες που έχετε. Τα πρόσωπα τα οποία δεν τα υποδέχονται και δεν αναγνωρίζονται ε, ως πρόσφυγες. Πού πρέπει να πάνε, πού επαναπατρίζονται, παραμένουν σε αυτή τη χώρα ή υπάρχουν κάποιες συμφωνίες με τις χώρες οι οποίες υποδέχονται τα πρόσωπα αυτά για να τα προσανατολίσουν σωστότερα. Τώρα για τη διαχείριση αυτών των μονάδων υποδοχής των τροφίμων. Κοιτάξτε, ξέρετε ότι στην Ρώμη υπάρχει ένα ολόκληρο σύστημα για τους πρόσφυγες, το οποίο συμμετέχει η μαφία ουσιαστικά ε, και πολλοί πέφτουν θύματα εκμετάλλευσης. Πώς θα ελέγξετε λοιπόν τις οργανώσεις οι οποίες διαχειρίζονται αυτά τα, τους χώρους υποδοχής. Ευχαριστώ πολύ, Σεσίλ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όταν άκουσα με προσοχή τις δύο παρουσιάσεις, πρόσεξα ότι ε, δεν επιμείνατε στην ανάγκη για βοήθεια επιτόπου και ιδιαίτερα στα στρατόπεδα των προσφύγων. Θα πρέπει λοιπόν τα κράτη-μέλη να είναι προσεκτικά σε σχέση με τον τρόπο που χρησιμοποιούν τα χρήματα των φορολογουμένων. Αλλά θα ήθελα να μπορέσουμε να βοηθήσουμε ε, τα παιδιά ε, εκεί που βρίσκονται μέσω της δημιουργίας σχολικών μονάδων. Μιλήσατε για την Σουηδία και εγώ είμαι Σουηδή και πράγματι εμείς στη Σουηδία έχουμε υποδεχθεί τους περισσότερους ε, και όλοι λένε ότι είμαστε οι καλοί μαθητές αλλά ξέρετε τι προβλήματα έχουμε να αντιμετωπίσουμε σε επίπεδο ενσωμάτωσης και εμείς έχουμε ανάγκη από βοήθεια και οικονομική βοήθεια για να καλύψουμε το κόστος των αναγκών που δημιουργεί αυτό το κύμα των, της υποδοχής. Εγώ δεν ξέρω αν η Σουηδία είναι πράγματι καλός μαθητής. Η χώρα μου υποδέχεται τους Ιρακινούς και τους Σύρους που ήρθαν για λίγο υποτίθεται, αλλά οι οποίοι δεν θέλουν να επιστρέψουν στις χώρες τους, θέλουν να παραμείνουν στην Σουηδία. Και γι' αυτό θα πρέπει να μην μας λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση αν θα πρέπει να υποδεχόμεθα ή όχι ε, τους πρόσφυγες. Το θέμα είναι τι γίνεται με αυτούς. Σίγουρα κάθε χώρα θα πρέπει να ορίζει μια συγκεκριμένη ποσόστοση, αλλά το θέμα είναι και από εκεί και πέρα τι γίνεται. Άκουσα με προσοχή επίσης και αυτά τα οποία είπαν οι εκπρόσωποι της Frontex και γνωρίζω ότι οι εγκληματίες βάζουν μέσα σε ταχύπλοα εκατοντάδες κόσμου και νομίζω ότι εκεί πρέπει να θέψουμε την προσοχή μας και το Frontex πρέπει να ασχοληθεί ακριβώς όχι ουσιαστικά με τους μετανάστες αλλά με αυτούς οι οποίοι περνούν τον κόσμο, τους παράνομους αυτούς που δήθεν διευκολύνουν τους πρόσφυγες. Κύριε Γιουρέκ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα, συγχαρητήρια στην ύπατη αρμοστία για το έργο της. Το γνωρίζω και εγώ το έργο σας στο ΜΑΝ, στη Βηρητό. Είναι μια πολύ σημαντική δουλειά, πράγματι. Και πιστεύω ότι πρέπει να υπογραμμίσουμε ιδιαίτερα τη συνεργασία μεταξύ των χωρών και με τις χώρες που έχουν πρόσφυγες που φεύγουν από τον πόλεμο, από τη Συρία για παράδειγμα. Προς όφελος των ανθρώπων αυτών θα πρέπει να ξέρουμε ότι οι περισσότεροι από αυτούς θέλουν να επιστρέψουν στη χώρα τους, στη χώρα από την οποία αναγκάστηκαν κάποια στιγμή να φύγουν. Άρα πρέπει να τους βοηθήσουμε διασφαλίζοντάς τους ότι επιστρέφοντας θα μπορέσουν να συνεχίσουν τη ζωή τους κανονικά. Πώς χρησιμοποιούμε τα χρήματα που έχουμε στη διάθεσή μας. Στο Λίβανο μας είπαν ότι δεν υπάρχει αναλογία σωστή στα χρήματα που παίρνουν εκείνοι κατά αναλογία με άλλες χώρες που υποδέχονται πρόσφυγες, ενώ βρίσκονται δίπλα στην μεγαλύτερη σημερινή κρίση εκείνη της Συρίας. Υπάρχουν μεγάλες ροές, πολύ σημαντικές προσφύγων που φεύγουν από τη χώρα τους. Το είπε και αναγκόμες πριν από λίγο. Είναι ανήκουστα αυτή η κατάσταση, χωρίς προηγούμενο. Ο αριθμός των προσφύγων είναι πάνω από το 30% του συνολικού πληθυσμού της χώρας. Γι' αυτό λοιπόν σας αθαρρύνω να αναθεωρήσετε τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η κατανομή των κονδυλίων. Να δώσετε περισσότερα χρήματα εκεί. Με αυτό τον τρόπο βοηθάμε και τους αυτούς μας. Δεν θα χρειάζεται μετά να υποδεχόμαστε στις χώρες μας τους πρόσφυγες αυτούς. Μπορούμε να περιμένουμε ότι όταν λήξει ο πόλεμος θα επιστρέψουν οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι ζουν σε καταβλισμούς, αλλά μετά να μπορούν τα χρήματα αυτά να τα χρησιμοποιήσουν για παράδειγμα να αγοράσουν ένα σπίτι στις χώρες τους αντί να τα ξοδεύουν σε εμά για να έρθουν σε εμά. Ο κύριος έχει λόγο. Ή κυρία Πάγιο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Είμαι από τη Σουηδία κι εγώ. Και στο Σουηδικό Κοινοβούλιο υπάρχει μια μεγάλη πλειοψηφία που υποστηρίζει την ανθρωπιστική υποδοχή των προσφύγων. Το λέω αυτό για να φανεί η διαφορά με την προηγούμενη Σουδέζα που μίλησε. Πολλοί το είπαν ότι πρέπει να βοηθήσουμε περισσότερο τα παιδιά στους καταβλισμούς προσφύγων, στο Λίβανο για παράδειγμα, αλλά όχι μόνο εκεί και αλλού, ακόμα και στη δικιά μου τη χώρα, εκεί όπου υποδεχόμαστε πρόσφυγες πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη σημασία στα παιδιά και τελείως θα χάσουμε μια γενιά αν δεν το κάνουμε. Πρέπει οπωσδήποτε τα παιδιά αυτά να έχουν μια προοπτική στη ζωή τους. Δεν είναι μόνο το θέμα της εκπαίδευσης, του σχολείου, αλλά και η ψυχολογική στήριξη, η κοινωνική βοήθεια. Τα παιδιά αυτά θα χρειαστούν πολλή βοήθεια στο μέλλον για να σωθούν, για να μην αποτελέσουν μέρος μιας χαμένης γενιάς. Είναι αλήθεια ότι υπάρχουν άνθρωποι που δεν θέλουν να επιστρέψουν στις χώρες τους, άλλοι όμως θέλουν να επιστρέψουν στις χώρες τους. Ορισμένοι όταν απορριφθεί το αίτημά τους για άσυλο, αποφασίζουν να γυρίσουν πίσω. Με πολλές δυσκολίες όμως. Στα στατιστικά στοιχεία δεν βλέπουμε τελικά ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι επιστρέφουν εθελοντικά. Βλέπουμε συνήθως αυτοί οι οποίοι απελάσσονται, που διώχνονται με το ζόρι και μάλιστα με πολύ ταπεινωτικό τρόπο. Αυτές λοιπόν οι απελάσεις είναι κάτι που συζητάμε πιο συχνά και όχι την εθελοντική επιστροφή, θέλω να πω στα μέσα ενημέρωσης. Αυτά διαβάζουμε κυρίως. Διαβάζουμε και αυτούς οι οποίοι δεν θέλουν να επιστρέψουν και επιστρέφουν με το ζόρι. Αλλά εγώ θέλω να ρωτήσω, αυτή την αναλογία τη γνωρίζετε, έχετε τέτοια στατιστικά στοιχεία για να μου πείτε πώς είναι αυτοί οι οποίοι απελάσσονται και πώς είναι αυτοί οι οποίοι επιστρέφουν στις χώρες τους σε θελοντική βάση ή και Σας ευχαριστώ όλους για τις εξαιρετικές ερωτήσεις σας. Αυτή την πέμπτη το απόγευμα έχουμε πάρα πολύ μεγάλο έργο να κάνουμε με την κοινή έκθεση για την μετανάστευση και είναι πολύ καλός πρόδρομος λοιπόν αυτή η συζήτηση, πάρα πολύ χρήσιμη. Και από την ε, τελευταία συνέντευξη του Συμβουλίου στη Ρίγα είχα την ε, εντύπωση ότι ε, είχα, την, είχα αποκομίσει μάλλον μία εντύπωση για το τι κάνουν τα κράτη-μέλη τι εντύπωση έχετε, δεδομένου μάλιστα ότι οι Αυστριακοί προσπαθούν αυτή τη στιγμή να ζητήσουν από τα κράτη-μέλη να αλλάξουν τη στάση τους απέναντι στην επανεγκατάσταση και δεδομένου ότι υπάρχουν κάποιες χώρες που είναι πάρα πολύ επιβαρημένες από ε, αυτή την αλλαγή από τους πρόσφυγες, η Ορδανία, η Τουρκία. Και να σας πω κιόλας ότι Υπάρχουν πολλά κρατημέλη και όχι μόνο η Αυστρία που έχουν μια παρόμοια άποψη. Εσείς βλέπετε κάποια τέτοια αλλαγή ή όχι. Τι εντύπωση αποκομίσατε από αυτές τις ε, συναντήσεις. Πώς υπάρχει επιθυμία για βελτίωση. Ποιος θέλει να αρχίσει. Εσείς κύριε Μούσελ. Θα θέλατε να απαντήσω τις δικές σας ερωτήσεις πρώτα ή τις ερωτήσεις των μελών. Αρχίστε πρώτα με τα μέλη μας και απαντήστε στη δική μου ερώτηση τελευταία. Πρώτη ερώτηση. Ε, μου κάνατε μία πάρα πολύ δύσκολη ερώτηση, το τι γίνεται δηλαδή εάν στα πλαίσια του προγράμματος επανεγκατάστασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης κάποιος ε, εισέλθει σε ένα κράτος της Βαλτικής για παράδειγμα και μετά από λίγους μήνες βρεθεί στη Γερμανία αν υπάρχει κάποιο είδους ε, συμβόλαιο με αυτούς τους ανθρώπους που επανεγκαθίστανται εάν του παίρνουμε από αυτά τα στρατόπεδα προσφύγων στην Ιορδανία, ε, για παράδειγμα, με την προϋπόθεση να μείνουν στη χώρα στην οποία θα επαναγκατασταθούν. Και ότι εάν σας βρούμε σε άλλη χώρα θα σας στείλουμε πίσω. Κάπως έτσι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε, μόνο έτσι. Και αυτό θα είναι και κάτι το οποίο θα παρακολουθούμε στα πλαίσια του πιλωτικού αυτού προγράμματος, δηλαδή τις δευτερογενείς μετακινήσεις όπως τις λέμε. πρέπει να παρακολουθήσουμε λίγο το σύστημα αρχικά και αρχικά πρέπει ο άνθρωπος αυτός να παραμείνει στη χώρα στην οποία θα επαναγκατασταθεί και μετά να εκτιμήσουμε την κατάσταση και να δούμε τι θα γίνει και αν μπορούμε να υποφεληθούμε από τη μετακίνησή του. Έπειτα ε, να σας πω, όσον αφορά τη δεύτερη ερώτηση, ότι είμαστε Έχουμε πλήρη επίγνωση για την κατάσταση στο Λίβανο, στην Τουρκία, στην Ιορδανία. Γι' αυτό και η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο υπαριθμόν ένα δονητής, ε, δωρητής στην περιοχή. Έχουμε διαθέσει πάρα πολλά κονδύλια για την σταθεροποίηση και βελτίωση της κατάστασης των προσφύγων, όμως είμαστε σίγουροι πως αυτό δεν φτάνει. Αν δείτε τι γίνεται με τη Συρία θα δείτε ότι την πρώτη χρονιά είχαμε 25.000 πρόσφυγες, τη δεύτερη 50, την τρίτη 100.000 πρόσφυγες. Υπάρχει γεωμετρική πρόοδος και όσο περισσότερο χρόνο αφιερώνεις στην κατάσταση στα στρατόπεδα προσφύγων, τόσο πιο πολύ απελπίζεσαι, γιατί βλέπεις ότι πραγματικά η κατάσταση είναι απελπιστική και σίγουρα χρειάζεται να γίνουν πάρα πολλά πράγματα και σε αυτό θέλουμε τη στήριξή σας. Το ζήτημα της Frontex τώρα. Ε, κυρία Χόλμαερ και τη στρατιωτική εκδοχή. Νομίζω δεν είναι δική μου αρμοδιότητα. Είμαι υπεύθυνο για την προστασία ε, των μεταναστών και όχι για τη στρατιωτική προστασία. Όμως έχετε δίκιο. Θα πρέπει να εξετάσουμε ένα τέτοιο ενδεχόμενο και να δούμε τι εμπειρίες αποκομίσαμε από την περίπτωση της Σομαλίας και ε, σίγουρα ε, είμαι, απόλυτα βέβαιος ότι αυτοί οι διακινητές πρέπει να αντιμετωπιστούν και ίσως με, στρατιωτικό, με στρατιωτικές μεθόδους. Και με ρωτήσατε και κάτι που εμπίπτει στις δικές μου αρμοδιότητες, η επαναγκατάσταση και για ορισμένα κράτη-μέλη τα οποία θέλουν να επιλέγουν τους ε, ανθρώπους που θα επαναγκατασταθούν. Εάν πραγματοποιηθεί αυτό το πιλωτικό πρόγραμμα θα υπάρχει λοιπόν ένας ε, λόγος ε, διανομής και θα λέμε για παράδειγμα η Γερμανία τόσους θα δεχτεί αλλά δεν θα υπάρχει επιλογή το, του ποιος θα πάει εκεί. Και φυσικά δεν θα επικεντρωθούμε μόνο στους ε, Σύριους, γιατί υπάρχουν κάποια κράτη-μέλη τα οποία θέλουν να βοηθήσουν ανθρώπους κάθε εθνικότητας και θα προσπαθήσουμε να είμαστε αντικειμενικοί, διότι όπως σας είπα στόχος μας ε, είναι να προσελκύσουμε όσο δυνατόν περισσότερα κράτη-μέλη στο πρόγραμμα αυτό. Και κυρία Σίπελ, συμφωνώ απόλυτα με τα σχόλιά σας. Καθήκον μας είναι να πάρουμε με το πλευρό μας ε, όλα τα κρατημέλη και σίγουρα υπάρχουν κάποιες ε, αντιρρήσεις και σίγουρα υπάρχουν κάποια κρατημέλη τα οποία μέχρι τώρα δεν έχουν συμμετάσχει ποτέ σε τέτοιες ε, δραστηριότητες και θα χρησιμοποιήσουμε διάφορες οντού την ΕΑΣΟ για παράδειγμα, έτσι ώστε να βοηθήσουμε αυτές τις χώρες να αρχίσουν να συμμετέχουν σε, την, σε αυτά τα προγράμματα επανεγκατάστασης. Τώρα η κυρία Κίνγκε έφυγε, δυστυχώς, αλλά να σας πω ότι για το ζήτημα της επιστροφής, ε, φυσικά και δεν ε, στέλνουμε κανέναν πίσω σε επικίνδυνη περιοχή, δεν θα στέλναμε κανέναν πίσω στη Λιβύη, αλλά υπάρχουν περιπτώσεις όπου η αίτηση κάποιου για άσυλο έχει απορριφθεί και εκεί προσπαθούμε να εξισορροπήσουμε ε, την κατάσταση και να εξετάσουμε το ενδεχόμενο μιας εθελοντική επιστροφής. Αν δεν κάνω λάθος τα νούμερα, το 30% των επιστροφών είναι εθελοντικέ και οι υπόλοιπες όχι. Το ενδιαφέρον όμως είναι ότι υπάρχει μία θετική τάση και αυτή είναι η τάση της αύξησης των εθελοντικών επιστροφών. Τώρα, όσο για τη Σουηδία. Να σας πω ότι αν όλα τα κράτη έκαναν το ίδιο πράγμα με τη Σουηδία, τότε η κατάσταση θα ήταν πάρα πολύ καλύτερη και θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε ακόμα περισσότερους ανθρώπους να επαναγκατασταθούν στην Ευρώπη. Κυρία Βίνμπεργκ, συνεχίζουμε στη Σουηδία. Με ρωτήσατε τι κάνουμε για αυτούς τους λαθρεμπόρους, τους σωματέμπους. Στις 20 Μαρτίου ημερομηνία προς επιβεβαίωση από την Ευρωπόλ, θα αρχίσει μια νέα επιχείρηση, Jot Mare είναι το όνομά της, όπου θα προσπαθήσουμε να καταπολεμήσουμε αυτούς τους διακινητές και θα πραγματοποιηθεί η επιχείρηση αυτή τους επόμενους μήνες. Είναι μια κύρια προτεραιότητά μας, αλλά δεν είναι μόνη της. Αποτελεί μέρος μιας δέσμης μέτρων. Τέλος. Ερώτηση δική σας κύριε Πρόεδρε. Κάτι κινείται πιστεύω στο Συμβούλιο και παρατηρώ μια θετική αντίδραση με αυτήν την πρωτοβουλία του, το Safe Lives. Ναι, λέει ο Πρόεδρος, κίνηση υπήρχε, αλλά δεν ήταν σωστή κίνηση. Μου φαίνεται πως ε, κάναμε κύκλους εσείς δηλαδή που νομίζετε πως πήγαινε αυτή η κίνηση. Νομίζω πως ε, δεν ήταν ένα κάθετο όχι στο πιλωτικό πρόγραμμα. Ναι, ναι, ξέρω, ξέρω, είστε δημόσιοι υπάλληλοι, κάπως έτσι μιλάτε, πείτε μου κι άλλα. Ναι, το σχέδιο λοιπόν είναι να πάμε στο επόμενο Συμβούλιο του Ιουνίου με το πιλωτικό πρόγραμμα ε, και αυτόν τον ε, λόγο της διανομής και να πιάσουμε τους υπουργού έναν έναν και να τους πούμε εσείς πόσους θέλετε να πάρετε, πόσους δέχεστε και αν δεν θέλετε να δεχτείτε αυτόν τον αριθμό που σας προτείνουμε, πείτε μας γιατί και πείτε μας τι θα κάνετε ανταυτού. Θα δώσετε χρήματα για το Λίβανο, για την Τουρκία, αντί, για, αντί να δεχτείτε πρόσφυγες. Και αν δεν συμμετέχετε στο πρόγραμμα, τι θα κάνετε. Αυτό είναι το σκεπτικό μας, αλλά θα δούμε αν θα πετύχει. Εσείς όμως να συνεχίσετε να ασκείτε πίεση, γιατί αυτό θα μας βοηθήσει. Ήθελα όχι μόνο να πληροφορηθώ εγώ, αλλά να πληροφορηθούν και τα μέλη μας για το αν υπάρχει κάποια θετική αντίδραση στην Αυστριακή Πρωτοβουλία. Γιατί σίγουρα υπάρχουν καλές πρακτικές από τις οποίες θα μπορούσαμε να διδαχθούμε και είναι παραδείγματα προς μίμηση, αλλά να συνεχίσετε να μας κρατάτε ενήμερους και εμείς θα συνεχίσουμε να ασκούμε πίεση. Καλώς. Η Φιλίπα τώρα. Thank Σας ευχαριστώ πολύ. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο. Υπήρξαν πολλές ερωτήσεις για τα στρατόπεδα των προσφύγων και ιδιαίτερα για την κατάσταση των παιδιών και την εκπαίδευση στα στρατόπεδα αυτά. Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα αυτό και το παραδεχόμαστε. Είναι βέβαια και προτεραιότητα για την αρμοστία σε συνεργασία με τη UNICEF, σε συνεργασία με ΜΚΙΟ, να προσπαθούμε να παρέχουμε εκπαιδευτικές υπηρεσίες στα παιδιά οι ανάγκες είναι τεράστιες. Στη Συρία ήδη οι ανάγκες είναι πραγματικά τεράστιες. Ε, παίρνουμε βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από μεμονωμένους χώρες, από όλο τον κόσμο. Παρ' όλα αυτά όμως αυτό δεν αρκεί για να μπορέσουμε να καλύψουμε ε, τις ε, ε, ανάγκες αυτών των ανθρώπων. Ξέρετε ότι έχουμε και επιπλέον καταστάσεις περίεργες όπως στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, στο Νότιο Σουδάν, έχουμε την αυξανόμενη κρίση στην Ιγυρία και έχουμε και το θέμα της Λιβύης. Είναι κάτι που μας ανησυχεί ιδιαίτερα η κατάσταση εκεί. Ξέρετε ότι ε, όλοι οι εκπρόσωποι των διεθνών οργανώσεων και ΜΚΟ έπρεπε να εγκαταλείψουν τη Λιβύη και έχουμε κάποιους βέβαια εκεί Λιβύους οι οποίοι εργάζονται στις υπηρεσίες μας αλλά και αυτοί μπορεί να χρειαστεί να μετακινηθούν γιατί η κατάσταση χειροτερεύει. Αυτές είναι καταστάσεις τις οποίες προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε αλλά η ύπατη αρμοστία έχει ήδη επαναλάβει ότι αυτό το οποίο απαιτείται είναι μια πολιτική λύση. Οι ανθρωπιστικοί παράγοντες κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους αλλά δεν μπορούν να λύσουν αυτό το πρόβλημα. Η πολιτική. Πολλοί από αυτού βρίσκονται εδώ. Είναι πολιτικό πάντω το θέμα και απαιτείται πολιτική λύση για την επίλυση αυτών των προκλήσεων. έτσι ώστε να μπορέσουμε να ελαφρύνουμε λίγο τα προβλήματα των ανθρώπων αυτών. Υπήρξαν και άλλα θέματα που αφορούν την επανεγκατάσταση ο συνάδελφός μου αναφέρθηκε σε κάποια από αυτά. Η αρχική διαδικασία είναι κάτι το οποίο μας έχει απασχολήσει. Προσπαθούμε εμείς καταρχάς να ταυτοποιήσουμε τα πρόσωπα που είναι στην κατηγορία της επανεγκατάστασης, αλλά οι περισσότερες από τις χώρες ε, εμπλέκονται στη διαδικασία επιλογής, μόνο σε πολύ λίγες περιπτώσεις που ε, εξετάζονται τα θέματα αυτά γενικά. Πάντως οι χώρες υποδοχής ε, προφανώς και έχουν λόγο στη διαδικασία και είναι πάρα πολύ λογικό αυτό. Τώρα σχετικά με τη δήλωσή μου και ε, ότι εννοούσα όταν αναφέρθηκα στην επιχείρηση τρίτων και στην εμβέλεια και τον στόχο της επιχείρησης τρίτων. Φυσικά, εμείς είμαστε υπέρ της συμπερίληψης της έρευνας και διάσωσης στον κανονισμό αυτό. Αυτό το οποίο θα ήθελα να πω είναι ότι δεν είναι ο πρωταρχικός στόχος του τρίτων, αυτό της επιχείρησης τρίτων. Το είπε και ο κύριος Μιουσέλ. Υπάρχει σαν στόχος και τους τελευταίους μήνες έχουν πάρει μέρος σε πολλές τέτοιες προσπάθειες διάσωσης, αλλά οι δυνατότητες τις οποίες έχουν είναι περιορισμένες. Τώρα για την άνηση κατανομή στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτών που ζητούν άσυλο. Και γιατί κάποιοι που φτάνουν σε μία χώρα ε, δεν ε, ζητούν άσυλο αλλά επιδιώκουν να πάνε σε άλλη χώρα. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο προσπαθούμε να λύσουμε. Είναι κάποια νέα τακτική αν θέλετε. Οι άνθρωποι κινούνται για διάφορους λόγους. Κάποιοι από τους λόγους αυτούς ελέγχονται από μας. Ε, υπάρχει διαφορετική εφαρμογή του συστήματος ασύλου στις διάφορες χώρες και φυσικά οι συνθήκες υποδοχής είναι εντελώς διαφορετικές αυτό μας το λένε όλοι οι πρόσφυγες, μας είπαν ότι σε ορισμένες χώρες δεν είχαν συστήματα υποδοχής. Λοιπόν, γι' αυτό το λόγο χρειάστηκε να προσπαθήσουν να πάνε αλλού. Υπάρχει το θέμα της οικογενειακής επανένωσης. Ε, θα προσπαθήσουν να πάνε σε χώρες τις οποίες έχουν μέλη οικογένειας, ακόμα και αν είναι μακρινά μέλη οικογένειας. Το γεγονός ότι έχουν κάποιους συγγενείς και κάποιες κοινότητες στις χώρες αυτές τους βοηθά και μπορεί να βοηθήσει και την ε, επανεγκατάστασή τους και την ολοκλήρωσή τους. Δεν είναι κάτι το αρνητικό υποχρεωτικά δηλαδή γι' αυτό. Λοιπόν δεν έχω κάτι άλλο να προσθέσω εδώ, ξέρω ότι δεν υπάρχει και πάρα πολύ χρόνος, αυτά. Είναι αλήθεια ότι είναι πάρα πολλά τα θέματα και θα επανέλθετε θα ζητήσω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κλείσει τη συζήτηση αυτή και να μας πείτε εσείς η Επιτροπή το πότε θα ε, ολοκληρωθεί η πιλωτική φάση. Ναι. Πρόκειται να έχουμε συνάντηση για την ε, μετεγκατάσταση και την επανεγκατάσταση όσο γίνεται πιο γρήγορα θα συζητήσουν οι επίτροποι την επόμενη εβδομάδα δηλαδή για την ε, ατζέντα όσον αφορά την μετανάστευση. Επίσης ετοιμάζουμε ήδη έγγραφο με την κλίδα κατανομής και περιμένουμε το πράσινο φως από τους επιτρόπους. Όταν θα το έχουμε, τότε τον Απρίλιο θα υπάρξει πλήρης ε, συνάντηση για να καταλήξουμε από κοινού και να μπορέσουμε μετά να πιέσουμε και τους υπουργούς να αποφασίσουν. Αυτό είναι το χρονοδιάγραμμα. Ωραία, λέει ο Πρόεδρος, έτσι κλείνει η συζήτηση. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ λοιπόν. Αγαπητοί συνάδελφοι, τώρα περνάμε στο επόμενο σημείο, σημείο 9. Πρόκειται για ένα θέμα που έχει να κάνει με τη στρατηγική μας εσωτερικής ασφάλειας. Πρόκειται για την σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για το κυβερνοέγκλημα. Η νομική υπηρεσία είναι εδώ για τη σύμβαση αυτή μετά από αίτημα της Επιτροπής μας όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις για ένα επιπλέον πρωτόκολλο όσον αφορά την πρόσβαση σε δεδομένα τα οποία είναι αποθηκευμένα σε υπολογιστή που βρίσκεται σε διαφορετική δικαιοδοσία. Και ιδιαίτερα για το θέμα του δικαιώματος και της αρμοδιότητας μάλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε διαπραγμάτευση. Ο κύριος Λουκάξη από την νομική υπηρεσία είναι εδώ. Σωστά. Είναι εδώ. Είναι εδώ ο κύριος Λουκάξη. Α, ξεχνάω ότι αριστερά κάθεται η νομική υπηρεσία και εγώ κοιτάω δεξιά μου πάντα. Γι' αυτό δεν σας είχα δει, συγγνώμη. Έλεγα λοιπόν ότι η Ιταλική Προεδρία πρώτα θέσαμε το ζήτημα αυτό της στρατηγικής μας για την ασφάλεια και ζητήσαμε γνωμοδότηση από την νομική υπηρεσία. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Αξιότιμοι Ευρωβουλευτές. Το Δεκέμβριο που μας πέρασε, η νομική υπηρεσία έλαβε έτοιμα για γνωμοδότηση όσον αφορά τη σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για το κυβερνάγκλημα. Πιο συγκεκριμένα, για τις εργασίες του Συμβουλίου της Ευρώπης όσον αφορά την παράταση μονομερής ε, διασυνοριακής πρόσβασης σε δεδομένα τα οποία είναι αποθηκευμένα σε υπολογιστή που βρίσκεται σε διαφορετική δικαιοδοσία. Δύο είναι τα ζητήματα. Πρώτον, ποια είναι η φύση της αρμοδιότητας Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα αυτό και δεύτερον, η προτινόμενη επέκταση είναι συμβατή με το ενωσιακό δίκαιο Εξετάσαμε λοιπόν τις εργασίες του Συμβουλίου της Ευρώπης βασιζόμενοι στα έγγραφα που είχαμε στη διάθεσή μας και καταλήξαμε ότι το υλικό που έχουμε στη διάθεσή μας είναι μόνο μερικό. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία βέβαια ότι αξίζει να μελετήσουμε πολύ περισσότερο το θέμα όσο προχωρούν και οι εργασίες στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Επιτρέψτε μου να σας πω δύο λόγια για την ίδια τη σύμβαση πρώτα. Πρόκειται για μια σύμβαση η οποία υπογράφηκε από όλες τις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από κάποιες ε, άλλες χώρες του Συμβουλίου της Ευρώπης. Καθώς και από άλλες χώρες εκτός Ηνωμένε Πολιτείε και η Ιαπωνία, για παράδειγμα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αποτελεί μέρο τη σύμβαση. Η σύμβαση λοιπόν έχει τρει ε, στόχους. Πρώτον, να αναρμονίσει το ουσιαστικό ποινικό δίκαιο όσον αφορά τα δικήματα στον κυβερνοχώρο. Δεύτερον, για ποινικό ναι, δικαστικό δίκαιο και τρίτον να δημιουργήσει ένα καθεστώς για τη διεθνή συνεργασία. Το θέμα που τίθεται αφορά την τρίτη αυτή κατηγορία, δηλαδή τη διεθνή συνεργασία. Η διάταξη αυτή έχει να κάνει με τη διασυνοριακή πρόσβαση σε στοιχεία υπολογιστή σε δύο περιπτώσεις. Όταν είναι δημόσια τα δεδομένα και δεύτερον στην περίπτωση όπου τα δεδομένα βρίσκονται σε μία άλλη πλευρά, σε ένα άλλο μέρος και το μέρος το οποίο ερευνεί παίρνει νόμιμα και σε θελοντική βάση τη συνένεση κάποιου ο οποίος έχει την άδεια να αποκαλύψει δεδομένα. Θα έχετε διαπιστώσει ότι είναι θέμα εδαφικότητας. Οι ερευνητικές αρχές δεν πρέπει να ακολουθούν τον παραδοσιακό τρόπο της αμοιβαία αρρωγής. Μπορεί να επεκταθεί πάντως η βοήθεια από καιρού καιρό στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Προς το παρόν, τα σχέδια αυτά αποτελούν μόνο κάποιες ιδέες, τροφή προσκέψη και δεν πρόκειται για ένα συγκεκριμένο νομικό κείμενο. Μετά από χρόνια λοιπόν προβληματισμού και συζητήσεων, το Συμβούλιο της Ευρώπης με την Επιτροπή του για τη Σύμβαση για τον Κυβερνοχώρο αποφάσισε το, αποφάσισε το Δεκέμβριο που μας πέρασε και στα πλαίσια των διαπραγματεύσεων για το πρωτόκολλο της επέκτασης ότι δεν είναι εφικτό. Αλλά η Επιτροπή αποφάσισε επίσης να ξαναδεί το θέμα του κατά πόσο είναι εφικτό ένα τέτοιο πρωτόκολλο και αποφάσισε να δημιουργήσει μια ομάδα εργασία που θα ετοιμάσει κάποιες προτάσεις. Η εντολή τη ομάδα αυτή λύγει στα τέλη του 2016. Συνεπώς, το ζήτημα παραμένει επιτάπητο. Επιτρέψτε μου τώρα να έρθω στο θέμα της αρμοδιότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μας ζητήσατε να διευκρινίσουμε την φύση της αρμοδιότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την επέκταση της διασυνοριακής πρόσβασης. Εδώ υπάρχει το άρθρο 3, σημείο 2 της Συνθήκης Λειτουργίας Ευρωπαϊκής Ένωσης που λέει ότι η εξωτερική αρμοδιότητα και το θέμα των διεθνών συμφωνιών μπορεί να επηρεάσει και κάποιους κοινούς κανόνες πέρα από το στενό το πρώτο είναι λοιπόν να δούμε την ύπαρξη αυτής της ευρωπαϊκής αρμοδιότητας. Αυτή υπάρχει. Η σύμβαση έχει να κάνει με την αναρμόνιση του ουσιαστικού ποινικού δικαίου για το εγκλήμα. Έχει αρμοδιότητα η Ευρωπαϊκή Ένωση σύμφωνα με τις συνθήκες από αυτού και έχει ασκήσει την αρμοδιότητα αυτή εγκρίνοντας οδηγία το 2013 για επιθέσεις σε σχέση με συστήματα η σύμβαση επίσης αφορά και τη διεθνή συνεργασία μεταξύ των αρχών επιβολής του νόμου για την καταπολέμηση του κυβερνοχώρου και έχει αρμοδιότητα να προβεί σε μέτρα σχετικά με τη, τη συλλογή, συγγνώμη, την αποθήκευση, την επεξεργασία, την ανάλυση και την ανταλλαγή σχετικών δεδομένων στα πλαίσια της αστυνομικής συνεργασίας. Έχει ασκήσει το δικαίωμά της αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση, την αρμοδιότητα της αυτή, το 2006 με απόφαση πλαίσιο που απλοποιεί την ανταλλαγή πληροφοριών και μυστικών πληροφοριών μεταξύ αρχών επιβολής του νόμου των χωρών μελών. Μπορούμε να συμπεράνουμε λοιπόν ότι υπάρχει αυτή η εξωτερική αρμοδιότητα στον τομέα αυτό καταπολέμησης ε, εγκλημάτων χώρου. Το δεύτερο θέμα είναι να αναλύσουμε τη φύση της αρμοδιότητας αυτής. Είναι αποκλειστική ή είναι επιμερισμένη. Και το σκοπό της ανάλυσης αυτής πρέπει να δούμε ποιοι τομείς καλύπτονται από τους ευρωπαϊκούς αυτούς κανόνες. Πρέπει επίσης να συγκρίνουμε τις μελλοντικέ εξελίξεις, την φύση τους και το περιεχόμενό τους. Όπως είπα, η προπόθεση που πρέπει εδώ να αξιολογήσουμε είναι κατά πόσο η εν λόγω συμφωνία μπορεί να επηρεάσει τους κοινούς ευρωπαϊκούς κανόνες ή να τροποποιήσει το πεδίο εφαρμογή τους. Προσπαθήσαμε λοιπόν να το εκτιμήσουμε αυτό γενικά. Δεν χρειάζεται απόλυτη σύμπτωση ανάμεσα στους τομείς που καλύπτονται από το Ευρωπαϊκό Δίκαιο και τις υποχρεώσεις μας σε διεθνές επίπεδο. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε για αντίφαση μεταξύ των δύο. Μπορεί αυτό βέβαια να μην είναι σαφές, αλλά σε πρόσφατες αποφάσεις του δικαστηρίου που έχουν να κάνουν με απαγωγές παιδιών και τη σύμβαση της Χάγης, πολλές χώρες είπαν ότι θέλουν πιο περιοριστική ερμηνεία της αποκλειστικής ευρωπαϊκής αρμοδιότητας. Το δικαστήριο όμως συμφώνησε με τα επιχειρήματα του Κοινοβουλίου και μάλλον έδωσε ευρεία ερμηνεία της αρμοδιότητας αυτής. Συνεπώς η δικιά μας ανάλυση βασίζεται σε αυτή την περίπτωση. Δεν θα σας δώσω λεπτομέρειες και σημεία αναφοράς, αλλά ε, κάναμε την ανάλυση μας ε, βάσει αυτών και καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι οι διατάξεις του κοινοτικού δικαίου καλύπτουν σε ένα μεγάλο βαθμό τον τομέα που καλύπτει και η προτινόμενη σύμβαση και υπάρχει κίνδυνος οι ευρωπαϊκοί κανόνες να επηρεαστούν εφόσον επεκταθεί η διασυνοριακή πρόσβαση. Συνεπώς, η αποκλειστική εξωτερική αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δυνητικά ε, επηρεάζεται από την ε, από τέτοιες διεθνείς συμφωνίες για την επέκταση της διασυνοριακής πρόσβασης. Θα μου πείτε τώρα γιατί χρησιμοποιούμε ένα τόσο προσεκτικό λόγο όταν πρόκειται για δυνητικά αποκλειστική αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η απάντηση είναι ότι το Συμβούλιο της Ευρώπης δεν έχει καταλήξει σε ένα συγκεκριμένο κείμενο για τη διασυνοριακή αυτή πρόσβαση. Εξακολουθούν να υπάρχουν πολλοί παράγοντες άγνωστοι στην ανάλυση αυτή. Γι' αυτό θα ήταν προτιμότερο να συζητήσουμε για ε, ισχυρή δυνατότητα παρά για βεβαιότητα. Το δεύτερο τμήμα πάντως όσον αφορά την πρώτη ερώτηση έχει να κάνει με τις διαπραγματεύσεις. Εξακολουθεί να υπάρχει αβεβαιότητα. Πρέπει να δούμε πώς οι κανόνες αυτοί θα εφαρμοστούν και κατά πόσο τελικά θα υπάρξει διαπραγμάτευση επισχεδίου πρωτοκόλλου. Όταν έχει αποκλειστική αρμοδιότητα για διεθνή συμφωνία η Ευρωπαϊκή Ένωση, τι διαπραγματεύσει τι κάνει η Κομισιόν. Όσο για τον ρόλο των χωρών μελών, το δικαστήριο λέει ότι εφόσον εγκριθεί η απόφαση του Συμβουλίου που επιτρέπει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διαπραγματευτεί για ε, πολυμερείς ε, συμφωνίες, τότε αρχίζει η διαβούλευση σε διεθνέ επίπεδο. Αυτό δεν χρειάζεται αποχή από τα κράτη-μέλη, όμως ζητάει τουλάχιστον στενή συνεργασία μεταξύ των χωρών μελών και των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων για να διευκολυνθεί το καθήκον της Ευρωπαϊκής Ένωσης να διασφαλίσει την ε, συνοχή. Συμβατότητα με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο τώρα εφόσον επεκταθεί η διασυνοριακή πρόσβαση. Δεν ήμασταν σε θέση να απαντήσουμε στο ερώτημα αυτό, γιατί η δοκιμή που πρέπει να κάνουμε είναι εντελώ διαφορετική από τη δοκιμή που κάνουμε στην περίπτωση τη Ευρωπαϊκή αρμοδιότητα. Στην δεύτερη περίπτωση η ανάλυση αρχίζει συγκρίνοντας δύο τομείς. Αν υπάρχει συμβατότητα, τότε μπορούμε να συγκρίνουμε νομικές διατάξεις. Όπως είπε και το δικαστήριο, χρειάζονται επαρκείς πληροφορίες και όχι μόνο υποθέσεις σχετικά με μια συμφωνία και χρειάζεται ένα πολύ συγκεκριμένο και πλήρες πλαίσιο. Όμως, επί του παρόντος δεν υπάρχει τέτοιο πλαίσιο από πλευράς του Συμβουλίου της Ευρώπης. Αλλά όπω είπα, αυτό δεν επηρεάζει την απάντηση στην πρώτη ερώτησή σας για την αρμοδιότητα. Τα θέματα αρμοδιότητας και συμβατότητας δεν συνδέονται μεταξύ τους με την έννοια ότι η αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να είναι αποκλειστική ακόμα και αν το ε, πρωτόκολλο δεν αντιφάσκει με κανόνες τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Για να συνοψίσω, οι ανησυχίε σα για το θέμα αυτό επιβεβαιώνονται από την νομική μας ανάλυση. Πράγματι υπάρχει μεγάλη δυνατότητα η αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να είναι αποκλειστική. Από την άλλη πλευρά η συμβουλή μας είναι ότι είναι πάρα πολύ νωρίς να εξετάσουμε το θέμα της συμβατότητας με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Φυσικά οι νομικές υπηρεσίες είναι στη διάθεσή σας για να αναλύσουν το θέμα αυτό ιδιαίτερα όταν και εφόσον ένα σχέδιο πρωτοκόλλου για τη διασυνοριακή πρόσβαση αποκτήσει μια πιο συγκεκριμένη μορφή. Είμαι στη διάθεσή σας για να απαντήσω στις ερωτήσεις σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ σημαντική η συνεισφορά σας ε, γιατί υπάρχει και η σύμβαση ε, για την τρομοκρατία και είναι κάτι που στην Επιτροπή θα συζητηθεί το Μάρτιο. Υπάρχει και ένα πρόσθετο πρωτόκολλο, θα ασχοληθούμε με τους ξένους μαχητές, γι' αυτό λοιπόν η γνωμοδότηση αυτή είναι πάρα πολύ σημαντική για μας παρότι πιστεύετε πως θα πάρει καιρό να εκτιμηθούν όλες οι συνέπειες και η έκταση των επιπτώσεων. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για τη γενική στρατηγική της ασφάλειας. Θα ήθελα εδώ να συγχαρώ όλα τα μέλη που έχουν μείνει μέχρι τώρα και έχουν ακούσει με πάρα πολύ προσοχή τα όσα υπόθηκαν. Πολύ ενδιαφέροντα τα όσα ακούσαμε πράγματι. Και συγχαρητήρια ξανά σε όλους όσους εσάς που αντέξατε μέχρι τώρα. Είχαμε πολύ φορτωμένο πρόγραμμα σήμερα το απόγευμα. Η Μόνικα βλέπω πως ζητά το λόγο και είναι ανυπόμονη κιόλα. Δεν περίμενα να κάνει κανένα ερώτηση, αλλά βλέπω ότι η Μόνικα, εσύ θες να απευθύνει μια ερώτηση στις νομικές υπηρεσίες. Ναι. Καταρχάς, ε, μια διαπίστωση σήμερα το πρωί διατυπώθηκε η κατηγορία ότι τα κράτη-μέλη δεν ανταλλάσσουν μεταξύ τους δεδομένα και δεν τα μοιράζονται τα δεδομένα. Αυτή η κατηγορία νομίζω πως εδώ διαλύθηκε και μόλις αποδείχθηκε το αντίθετο, ότι τα κράτη-μέλη και ανταλλάσσουν μεταξύ τους δεδομένα και έχουν πάρα πολύ καλή συνεργασία και αν έχω καταλάβει καλά, υπάρχει μια πολύ, ε, ένας πολύ καλός διαχωρισμός, ότι τα κράτη-μέλη έχουν την ε, δικαιοδοσία να δρουν αυτόνομα μέχρι ε, να αποδειχθεί ότι δεν είναι αρμόδια. Από την ε, Επιτροπή αυτή, η αναρμοδιότητα, λοιπόν, μου φαίνεται κάπως περίεργη. Και μου κάνει τρομερή εντύπωση μάλιστα που αναφέρθηκε και το τι γίνεται στην ε, περίπτωση που κάποιο κράτος μέλος έχει διαφορετική άποψη από την Επιτροπή για το ποιος είναι αρμόδιος και ποιος είναι όχι. Και τι, τι, γίνεται σε αυτήν την περίπτωση, πώς θα βρεθεί λύση, πρέπει να προσφύγουμε στο δικαστήριο. Ναι, πράγματι, σε αυτή την περίπτωση δώσω την απάντηση στην ερώτησή σας. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος άλλος συνάδελφος ο οποίος έχει κάτι να ρωτήσει. Δώστε την απάντηση για να κλείσουμε με την υπόθεση. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να υπογραμμίσω εδώ ότι το σημείο εκκίνησης της κατάστασης είναι να σεβαστούν τα κράτη-μέλη αυτό το οποίο ζητάει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Συμβούλιο επιτρέπει τη διαπραγμάτευση μιας συμφωνίας. Δεν είμαστε κοντά σε αυτό, δεν υπάρχει μια τέτοια συμφωνία προς το παρόν, ούτε καν σε επίπεδο προτάσεως. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι υπάρχει εκκίνηση των διαπραγματεύσεων. Στα πλαίσια της ευρωπαϊκής νομολογίας υπάρχει ένα περιθώριο εδώ θα έλεγα το οποίο μπορεί να συμπληρωθεί με το συγκεκριμένο μόντους operandi, τους πραγματικούς κανόνες λειτουργίας. Λέγει το δικαστήριο ότι τα κράτη-μέλη δεν έχουν μια υποχρέωση διεύρυνσης των μέτρων αυτών, μπορούν όμως να πάρουν μέτρα. Πρέπει όμως να συνεργάζονται πάρα πολύ στενά με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Νομίζω λοιπόν ότι αυτό αφήνει ένα κάποιο περιθώριο δράσης για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη έτσι ώστε να προχωρήσουν σε κάποιες πρακτικές λύσεις ιδιαίτερα που στην συγκεκριμένη περίπτωση, στην περίπτωση δηλαδή των διασυνοριακών προσβάσεων μιλάμε για ερευνητικά μέτρα. Τα ερευνητικά μέτρα είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών όπως ε, γνωρίζετε και το δείχνει πολύ σωστά και η ε, ερώτησή σας. Κάποιες πρακτικές ε, λύσεις θα μπορούσαν να εμπλέξουν τα κράτη-μέλη, αλλά δυστυχώς αυτό δεν είναι θέμα αρμοδιότητας. Εάν οι αναλύσεις μας επιβεβαιωθούν στο μέλλον, θα υπάρξει μια πρόταση πρωτοκόλου συνεργασίας και τότε θα μπορέσουμε να πούμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ε, μια ε, αποκλειστική αρμοδιότητα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς την παρούσα φάση έχει τη δυνατότητα να διαπραγματευτεί τη συμφωνία και η ε, αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι απολύτως αποκλειστική. Στην πρακτική όμως τα κράτη-μέλη σίγουρα θα παίξουν κάποιο ρόλο στην διαπραγμάτευση της συμφωνίας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και τη Μόνικα για την εξαιρετική της ερώτηση. Συνάδελφοι, τελειώσαμε με το συγκεκριμένο θέμα. Ευχαριστώ την νομική υπηρεσία. Περνάω τώρα στο σημείο 10. Υπάρχει και τέτοιο. Και έχουμε τώρα την διαδικασία απάντησης στην Επιτροπή της κυρίας Γκαρντίνη. Μια ανταλλαγή απόψεων λοιπόν σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού. Στις 29 Οκτωβρίου η Αλιζαμπέτα Γκαρντίνη απέστειλε μία επιστολή για την εφαρμογή της, προ... της οδηγίας προσωρινής προστασίας. Απαντήθη και η ερώτηση αλλά όχι στον απαιτούμενο χρόνο των έξι εβδομάδων και ζητάμε λοιπόν τώρα λεπτομέρειες για την απάντηση αυτή. Η κυρία Γκαρντίνη είναι εδώ. Θα πρέπει να αρχίσω να ρωτάω πρώτα αν είναι εδώ οι ενδιαφερόμενοι πριν ξεκινήσει η συζήτηση. Υπάρχει και μία ερώτηση για την ε, ε, σύμβαση της Βουδαπέστης, πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Έπρεπε να τα πω νωρίτερα. Ζητώ συναδελφοί συγγνώμη, δεν τα προγραμμάτισα καλά, ζητώ συγγνώμη. Είναι πέντε παρατέταρτο, είναι πέμπτη απόγευμα. Ε, και τι να κάνουμε εδώ είμαστε. Όλοι καλοί είναι εδώ. Δεν ξέρω τι θα κάνουμε. Κοιτάξτε, αν αρχίσετε να φεύγετε όλοι, δεν ξέρω τι θα γίνει. Θα πρέπει να πάρουν κάποιο βραβείο η Μόνικα και ο Κοέλιο για την παραμονή τους εδώ. Δύο παρατηρήσεις για όποιους μας βλέπουν στο διαδίκτυο. Καταρχάς είχαμε πάρα πολλά θέματα σήμερα. Και δεύτερον, αν κάποιος λοιπόν επαναλαμβάνω παρακολουθεί, μέσα σε μία ώρα πήγαμε από τη Συρία και το Λίβανο, φτάσαμε ε, στην διάσκεψη για το κυβερνοέγκλημα, την διάσκεψη της Βουδαπέστης. Αυτό δείχνει πόσα και διαφορετικά τεχνικά θέματα είναι αυτά τα οποία πρέπει να μας απασχολούν. Και αυτό ισχύει φυσικά και για το προσωπικό, όχι μόνο για μας. Τα πράγματα έχουν αλλάξει εδώ και κάποια χρόνια. Και περιμένουμε. Ε, αν διακόψω για λίγο δεν νομίζω ότι θα επιστρέψει μετά ακόμα να κάνω διακοπή. search party is going out, Έχουμε στείλει μια αποστολή αναζήτησης υπό την αιγίδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Καλή τύχη. Ευχαριστώ Μόνικα Χορμάγερ. Πραγματικά ψάχνουμε με αγωνία ένα επιπλέον μέλος. Κοιτάξτε, αυτό έτσι και είναι το τελευταίο θέμα. Μια ανακοίνωση όσο περιμένουμε την εισηγήτρια. η ανακοίνωση για την... Να πω ότι σήμερα στις 6 παρατέταρτο έχουμε μία συνάντηση με την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων. <laughs> ναι, ναι, θα πρέπει να πάω κι εγώ για την ε, συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, στην 3G2. Παρουσίαση λοιπόν για την ένταξη της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ε, Σύμβαση. Όποιος θέλει παρακαλώ να έρθει, ελάτε. Νομίζω θα έχει ενδιαφέρον και θα το εκτιμήσω δεόντως. 3G2 στις 6 παρατέταρτο. You ready? Are you ready, Mrs. Gardini? Don't worry, we're waiting for you, but it's it's not your fault. You were probably timing your entry, but we we had finished the other item earlier. Are you ready to go? I've, I've introduced. Είσαστε έτοιμοι ε, για να ξεκινήσετε. Εγώ παρουσίασα την προφορική σας ερώτηση. Έχετε το λόγο για να την θέσετε. Σύντομα παρακαλώ. Ήδη έκανα την εισαγωγή. και θα ζητήσω επίσης ε, και την γνώμη του κυρίου Μουσέλ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, ζητώ συγγνώμη, αλλά μου είχατε πει στις 5 και ξαφνικά μου είπαν ότι τελείωσαμε νωρίτερα. Δεν ήθελα να σας καθυστερήσω, ζητώ συγγνώμη. Είναι ένα θέμα το οποίο με ενδιαφέρει ιδιαίτερος, όπως και σε πολλούς άλλους συναδέλφους. θα πρέπει να γίνει μια συζήτηση στη Λίμπε για το θέμα αυτό. Εν τω μεταξύ υπήρξε απάντηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την οποία είδα και η οποία με εκπλήσει θα έλεγα λίγο. Γιατί εάν πράγματι θεωρήσουμε ότι η σημερινή κατάσταση κάτω από τις παρούσες και συνθήκες ε, και κάτω από τις μεταναστευτικές ροές ε, δεν είναι τόσο σημαντική υπόθεση και ότι μπορεί κανείς να τα τακτοποιήσει όλα αυτά και να καταθέσει αυτήν την οδηγία με κανονικό τρόπο τότε πού βρίσκεται το χρήσιμο σημείο, γιατί το μόνο σημείο στο οποίο περιλαμβάνει την απάντησή της ότι 100.000 Συρίοι έχουν ζητήσει άσυλο από τον Ιανουάριο του 2014. Δεν έχω τα τελευταία στοιχεία γιατί από ό,τι φαίνεται δεν έχουν συλλεγεί, δεν έχουν ανακοινωθεί επισήμως. Αλλά βλέπουμε τι έγινε στο 12, είχαμε 335.000 αιτήσει το 14.440 περίπου. Συνεπώς λοιπόν με μια συστηματική αύξηση από τον ένα χρόνο στον άλλο ε, βλέπουμε ότι έχει υπάρξει πάρα πολύ σημαντική αύξηση από τη Συρία. Ζούμε μια δραματική κατάσταση. Βλέπουμε ανθρώπινα όντα τα οποία προσπαθούν να ξεφύγουν από μια περιοχή στον κόσμο η οποία καίγεται και θυμίζω ότι και εμείς κάναμε λάθος εκεί όταν ε, πιστέψαμε ότι θα βοηθούσαμε τη δημοκρατία και δεν ακούσαμε αυτούς που μας προειδοποιούσαν ότι η κατάσταση στη χώρα ήταν πολύ πιο περίπλοκη από όσο ονομάζουμε. Εμείς από την Ιταλία είμαστε αρκετά κοντά στις ζώνες από τις οποίες έρχονται όλοι αυτοί οι διαθαλάσσεις Πραγματι ξέρετε ότι σιγά σιγά η Μισόγειος έχει αρχίσει να μετατρέπεται σε ένα νεκροταφείο χωρίς στέγη. Λοιπόν, και η γραφειοκρατική αυτή αντίληψη με εκπλήσει. Θα ήθελα λοιπόν η απάντηση αυτή η οποία όπως είπα καθυστέρησε είναι μια πρόχειρη απάντηση από μια υπηρεσία η οποία δεν έχει συνειδητοποιήσει πλήρως το πρόβλημα και η οποία απάντησε ε, έτσι γιατί ξέρει ότι θα έχουμε κι άλλες ευκαιρίες να προσπαθήσουμε να δώσουμε απαντήσεις αλλά όπως είπαμε η απάντηση δεν ήταν ε, πλήρης. Ελπίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορέσει να δώσει μια απάντηση πολύ πιο ανθρώπινη, μια απάντηση πληρέστερη. Δεν θέλω να μακρηγορήσω, αλλά αν δείτε εσείς τις εκθέσεις των ΜΚΟ, αν δείτε τις εκθέσεις αυτών που φροντίζουν αυτή την κατάσταση, αν δείτε τα στοιχεία των γιατρών χωρίς σύνορα για, τις, για τους καταθλιπτικούς, για τις αυτοκτονίες, για την πορνεία, βλέπουμε ότι έχουμε μια λιτανία ουσιαστικά ανθρώπινου δράματος και θα πρέπει να ασχοληθούμε επιτέλους με αυτό με πάρα πολύ σοβαρότερο τρόπο. Λοιπόν, ποιο είναι το κρίσιμο σημείο για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πότε η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει, εν περιπτώσει, να ασχοληθεί σοβαρά με το θέμα αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί να σας κοιτάξει στα μάτια και να σας απαντήσει γιατί είναι πίσω σας, αλλά είναι εδώ, έτοιμη να απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις. Γι' αυτό λοιπόν, παρακαλώ Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δώστε μας τη δική σας εκδοχή. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Είμαι κάπως προβληματισμένος από αυτή την παρέμβαση της κυρίας Ευρωβουλευτή. Γιατί η ερώτηση ήταν για την οδηγία, την προσωρινή προστασία και όχι για την ε, στην Ευρώπη και το τι κάνουμε γενικότερα. Γι' αυτό λοιπόν αναρωτιέμαι εάν θα μπορούσαμε να... Ε, η ερώτηση μάλλον ήταν αν μπορούσαμε να πυροδοτήσουμε αυτό το μηχανισμό προσωρινής προστασίας και η απάντηση είναι όχι γιατί προ το παρόν δεν μπορούμε να θέσουμε σε ισχύ την αντίστοιχη οδηγία διότι επεξεργαζόμαστε ακόμα τα πράγματα διότι ο αριθμό των Σύριων που φτάνει είναι ένας διαχειρίσιμο αριθμός και όπως είδαμε μετά το, την κρίση στο Κόσοβο λειτουργήσε το σύστημα ασύλου και δεν εξετάζουμε την κάθε αίτηση για άσυλο σε αίτηση ασύλου, δίνουμε σε όλους ένα βασικό δικαίωμα προστασίας και όποιος φτάνει στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση παίρνει ένα καθεστώς ε, πρόσφυγα. Σύμφωνα λοιπόν με το κεκτημένο για το άσυλο, λαμβάνουν οι πρόσφυγες αυτό το καθεστώ του πρόσφυγα. Υπάρχουν υποστηρικτικοί μηχανισμοί μέσω τη ΕΑΣΟ. Έχουμε κάποιους μηχανισμούς ε, συνδρομή στην Ιταλία, τη Βουλγαρία, την Κύπρο και είναι αντιμετωπίσιμη λοιπόν η κατάσταση από το σύστημα. Ο αριθμός είναι διαχειρισμός, Δεν χρειάζεται λοιπόν να ε, τεθεί σε ισχύ το σύστημα προσωρινής προστασίας. Επιπλέον να σας πω ότι ούτε η Ιταλία ζήτησε αυτό το, ε, την οδηγία προσωρινής προστασίας, ούτε η Ελλάδα. Γι' αυτό δεν θεωρούμε πως αυτό το στάδιο είναι αναγκαία η θέση ισχύ του μηχανισμού προσωρινής προστασίας. Και να παραπέμψω το αξιότιμο μέλος σας σε αυτά που συζητήσαμε νωρίτερα το απόγευμα, όπου θα βρει και τις απαντήσεις της. Σας ευχαριστώ. Θα θέλατε να επανέλθετε σε αυτή την απάντηση. Σύντομα παρακαλώ. Κατανοώ ότι η απάντηση που μου δίδεται είναι γραφειοκρατική. Έχω μπροστά μου μια Ευρώπη που δεν είναι ευέλικτη. Έχουν φύγει 2,5 εκατομμύρια άνθρωποι από τη Συρία και δεν έχουν φτάσει μαζικά εδώ γιατί μεσολαβεί μια θάλασσα. Αλλά τα εκατομμύρια αυτών που βρίσκονται από την άλλη πλευρά της θάλασσας ε, θέλουν να έρθουν. Πρέπει λοιπόν να υπάρξει ευελιξία, να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα το οποίο έχουμε μπροστά μας μόνο και μόνο γιατί δεν υπάρχει μια διόρυγα για να περάσουν απέναντι. Αν υπήρχε θα είχαν ήδη έρθει εδώ. Ε, αυτό λοιπόν δεν το κατανοούν οι Ευρωπαίοι πολίτες και λυπάμαι που είμαι εδώ και πιέζω λέγοντας ότι η Ευρώπη κρύβεται πίσω από γραφειοκρατικά εμπόδια αντί να κάνει ένα βήμα ποιότητας και να αντιμετωπίσει την ανθρώπινη και την πολιτική πλευρά του προβλήματος. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Είναι καλό που έχουμε τη δυνατότητα να ακούσουμε και τις δύο πλευρές. Η Κομισιόν απάντησε στα τεχνικά στοιχεία κλειδί και εσείς από την πλευρά σας είπατε ότι πρόκειται για μια γραφειοκρατική απάντηση. Βλέπετε ευρύτερα το θέμα. Ωραία, είχαμε έτσι μια ανοιχτή ανταλλαγή εδώ στην Επιτροπή μας. Το καταγράφουμε. Έγινε αυτό που ζητήσατε. Θα παρακολουθήσουμε τη συνέχεια. Σας ευχαριστούμε <laughs> πάντως που ήρθατε. Ευχαριστώ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την απάντησή της. Αγαπητοί συνάδελφοι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας σήμερα το απόγευμα. Είναι το τελευταίο θέμα που είχαμε για σήμερα στην σε διάταξη. Θα μετακινηθούμε τώρα. Θα πάμε στην 3G2 αίθουσα, ώστε να δούμε το σημείο 13 για την πρόσβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Σύμβαση για την Προστασία Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Θεμελιωδών Ελευθεριών που θα αρχίσει στις 17 και 45, 6 παρατέταρτο δηλαδή, με την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων. Ελπίζω να έρθετε κι εσείς να βρεθούμε εκεί, υπό την Προεδρία της ΑΦΚΟ. Εντάξει, σας ευχαριστώ πολύ συνάδελφοι για όλη τη βδομάδα που ήσασταν μαζί μας. Αν δεν σας δω εκεί, σας αποχαιρετώ τώρα γιατί τελειώσαμε.